Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Θα μιλάω στα γερμανικά, λέει η πρόεδρος. Αυτό το κάνω για να χαροποιώ τους διερμηνείς, λέει η πρόεδρος, και για να τους δώσω δουλειά βεβαίως. Έχουμε συνέλθει σήμερα κυρίες και κύριοι για να ακούσουμε για να ακούσουμε τους τέσσερις υπουργούς της Ουγγαρίας για να ακούσουμε τα θέματα επί της παιδείας, του πολιτισμού, των κοινωνικών υποθέσεων, όλους αυτούς τους υπουργούς. Θα θέλαμε λοιπόν να πληροφορήσουμε για το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων μας, τι ακριβώς εξετάζουμε εμείς εδώ και τι θα πρέπει αυτοί, με τι θα πρέπει αυτοί να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια της Ογγρικής Προεδρίας. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ καλά. Είναι το, η ετικέτα όσον αφορά την ευρωπαϊκή κληρονομιά και για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει το Συμβούλιο να δουλέψει και, και βεβαίως εγώ έχουμε εδώ την πρώην Υπουργό πολιτισμού της Σλοβενίας η οποία είναι εισηγήτρια εδώ είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα αλλά παραλλήλως είναι και ένας μηχανισμός, ένα μηχάνημα το οποίο είναι εργαλείο που θα έχουμε στα χέρια μας για να μπορούμε πραγματικά πολύ καλύτερα να χρησιμοποιηθεί αυτό από τους νέους μας διότι ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με την βιομηχανία και τον πολιτισμό. Είναι όπως ξέρετε πάρα πολύ σημαντική η βιομηχανία του πολιτισμού αν θέλετε κατά τη διόρκεια της κρίσης καθότι μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε πάρα πολύ στο ΑΕΠ της χώρας, στο εθνικό, α, καθάριστο εθνικό προϊόν και ξέρετε πολύ ότι παίζει σημαντικό ρόλο για πολλούς εκ των συμπολιτών μας σαν ένας παράγων και εμπλουτισμού και ψυχαγωγίας αν θέλετε ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι φτάνουμε σε ένα τέρμινο, σε μια προθεσμία η οποία είναι καταλητική, πάρα πολύ σημαντική για την εκπόνηση αυτής τη εργασίας και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εργαζόμαστε εμεί με ιδιαίτερη στενή συνεργασία σε αυτά τα θέματα. Δεν θέλουμε κανένα να τον υποχρεώσουμε να κάνει κάτι που δεν θέλει, αλλά πρώτα θα θέλαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και στο Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να υποβάλουμε αυτά τα πράγματα σε όλους τους συναδέλφους για να δούμε πραγματικά τι θα αποφασιστεί και πώς πραγματικά τι γνώμονα θα έχουμε για την περαιτέρω εξέλιξη όλων αυτών. Πιστεύω πως κατά αυτόν τον τρόπο η... ψηφιακή μας δίνει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα, η ψηφιακή τεχνολογία, μας δίνει τη δυνατότητα να εργαστούμε πολύ περισσότερο και να κατορθώσουμε να βλέπουμε φιλμ, να βλέπουμε ταινίες δηλαδή, οι οποίες παλαιότερα δεν ήταν, ε, ήταν προνόμιο το λίγο, ενώ σήμερα έχουμε αυτή τη δυνατότητα όλοι μας από το σπίτι μας να δούμε και κατά αυτόν τον τρόπο ο πολιτισμός, η κουλτούρα να αναπτυχθεί περαιτέρω. Πιστεύουμε πραγματικά πως κατά αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερο πάμε προ, μπροστά και ευελπιστούμε πως κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ασχοληθούμε με τον πολιτισμικό χαρακτήρα χωρίς να ασχούμαστε μόνο, μόνο σε ένα και μόνο πράγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε προβλέψει αυτή την, την, ε, ε, την εισήγηση για να μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός είναι ο, αυτά ήθελα να σας πω εγώ εισαγωγικά και θα θέλαμε να σας ε, ε, ε, υποδεχθώ με πολύ χαρά και θα δώσουμε στον κύριο Ατσέλινγκ το λόγο, ο οποίος είναι υπουργό Αθλητισμού της Ουγγαρίας και βεβαίω θα του θέσετε ερωτήσεις οι οποίες είναι της αρμοδιότητας του. Και βεβαίω θα κάνετε το αυτό για τους άλλους υπουργούς που θα δεχτούμε αργότερα με τη σειρά τους εδώ. Μην διστάσετε λοιπόν να θέσετε τις ερωτήσεις οι οποίε θέλετε προς, προς τον Υπουργό και τους υπόλοιπους υπουργούς και εφόσον ένα ερώτημα δεν άπτεται του παρόντος Υπουργού μπορείτε να το κρατήσετε για αργότερα για, για αργότερα για τους υπόλοιπους υπουργούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ακρόαση. Ο κύριος Τιλατσένη, ο υπουργός, έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω κυρία Πρόεδρε η Ουγγαρία θα, είναι, θα υποστηρίσει την επιτροπή σας για όλα τα θέματα τα οποία αναφερθήκατε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, εγώ ως υπουργό ο οποίος ασχολούμαι με την αθλητισμό θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας εδώ ενώπιον της Επιτροπής σας. Ξέρετε, δύο παράγοντες επηρεάζουν την αθλητισμό στην αψινάψη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξέρετε ακριβώ πού πάνετε και υπάρχουν οι η απόφαση της, η ανακοίνωση της Κομισιόν της 19 η Γενουαρίου όσον αφορά τον αθλητισμό θα θέλαμε εμείς να οικοδομήσουμε μια εργασία με, το, με, την τριαρχία αν θέλετε Βέλγιο και ε, Ισπανία μια γερή βάση διότι θα πρέπει ε, να, η Ουγγαρία να παίξει το συντονιστή δηλαδή σε αυτό το θέμα θα πρέπει να υποστηρίξουμε μέτρα ή κίνητρα ή να κάνει προγράμματα εάν υπάρχει μια προστιθέμενη αξία ε, σε εθνικό επίπεδο για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό νομίζω πως λέγεται και επαναλαμβάνεται μέσα στο ανακοινωθέν της Κομισιόν για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης. Θα πρέπει να έχει μια προστιθέμενη ξύμια στην ΕΕ και θα πρέπει να ερχόμεθα με θέματα τα οποία παστής χρειάζεται όσον αφορά το αθλητισμό στην Ευρώπη. Καθότι αυτό το οποίο θέλουμε από τον αθλητισμό ακόμη περισσότερο είναι να από σήμερα μέχρι το 2014 υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει καθώ οποίε και οι αθλητικοί οργανισμοί να μα βοηθήσουν σε αυτό το θέμα, του ακουραστούμε και ό,τι άπτεται του αθλητισμού. Το Συμβούλιο σε αυτό το θέμα σε υψηλότερο επίπεδο έχει ασχοληθεί και η αποφάση του είναι πάρα πολύ σημαντική. Η σχέση μεταξύ Συμβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε τις απόψει των κρατών μελών για αυτό το θέμα και υπάρχουν πολλές ελπίδες για αυτό το θέμα του αθλητισμού εάν πραγματικά ε, ε, έρθει να προσθεθεί και να είναι σαφές, όπως είπε και ο Επίτροπος Βασιλείου, σε αυτή την ε, περίοδο της κρίσης. Νομίζω πως πραγματικά ο, από το 2014 και λοιπά θα είναι μόνιμες πολιτικές όπως είπε ο Επίτροπος Βασιλείου για αυτά τα θέματα όσον αφορά την νεότητα, την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μπαίνει ένα ολόκληρο πακέτο δηλαδή. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον αθλητισμό, να γίνει ένας κανονικός τομέα και ξέρετε ε, ο αθλητισμός καταρχήν είναι εθνικής αρμοδιότητας και η ΕΕ μπορεί να δράσει και είναι χρήσιμη και είναι επιθυμητέα αυτή η προσπάθεια που κάνει. Ο αθλητισμό μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, τους ομάδες, τους ε, ε, ε, θεατές κατά επίσης θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όρια τα οποία είναι κοινωνικά, οικονομικά ή άλλα. Είναι χωρί σύνολο αθλητισμό. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είναι πολύ γνωστό ότι κάθε κράτο μέλλον μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και σύμφωνα με τα συστατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε για το 10, η Κομισιό έχει δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ για τα project της κοινωνικής συνοχής, ε, της κοινωνικής ένταξης, του αθλητισμού, της νεολαίας καθώς επίσης ισότητα των φύλων και η υποστήριξη των ε, αναπήρων. Αυτή ήταν λοιπόν μια προπαρασκευαστική δραστηριότητα η οποία αναπτύχθηκε. 12 νέα σχέδια project έχουν λανσαριστεί αυτή τη χρονιά και η Ουγγαρία θα συμμετέχει, συμμετάσχει σε τέσσερα από αυτά τα προγράμματα. Ένα θα εστιαστεί πολύ, πολύ περισσότερο στο ντόπινγκ και ένα άλλο θα έχει σχέση για τον, ε, ε την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Αυτά είναι πρωτοβουλίες τις οποίες χαιρετίζουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε ένα πλαίσιο παρά τις αρχικές δυσκολίες. Τα κράτη-μέλη μπορούν ε, να εκμεταλλευτούν, ε, να χρησιμοποιήσουν τα δομικά ταμεία, τα ταμεία, διότι ο αθλητισμός είναι από τα νεότερα καθήκοντα αρμοδιότητες της ΕΕ που υπάρχει τελευταία και θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να δαπανούνται τα χρήματα στον αθλητισμό και να βελτιωθεί η, τα κονδύλια του προϋπολογισμού του αθλητισμού και νομίζω πως όλα τα μέλη αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα αυτής της Επιτροπής θα το κάνουν αυτό το πράγμα και ότι χρειαζόμαστε πολύ, πολλές περισσότερες πρωτοβουλίες για να δουλέψουμε μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Από τη Βελική Προεδρία μάθαμε ότι θα πρέπει να πάμε μπροστά με αυτές τις νέες πολιτικές και στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς επίσης με τη συνάντηση στο, στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Αθλητισμού και υπάρχει αυτή η ανακοίνωση της Κομισιόν με βάση την οποία το Συμβούλιο κάνει μια συνάντηση το Μάιο όπου θα υπάρχει ένα ψήφισμα γιατί Υπάρχουν ομάδες αθλητισμού οι οποίες εργάζονται επί των κειμένων τα οποία εκπονούνται εδώ στις Βρυξέλλες και θα είναι το πρώτο ε, δίκτυο α, θέλετε το οποίο θα θέσει όλες εκείνες τις προτεραιότητες που χρειάζονται για μένα. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή να υπάρχει εκ μέρους του Συμβουλίου ένα σχέδιο εκπονημένο για τις επόμενες προεδρίες οι οποίες έρχονται μετά από εμά. Για αυτή τη χρονιά και την επόμενη θα υπάρχουν δύο σημαντικά σημαντι γεγονότα τα οποία θα υπάρχουν. Πρώτο, η συν 23 και 23 Φεβρουαρίου οι Υπουργοί Αθλητισμών θα συνέλθουν. Επίσης θα υπάρξει ένα φόρουμ του αθλητισμού το οποίο θα συνέλθει και θα συμμετέχουν πολλές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη αθλητικές και θα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα, έρχονται από, θα συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ της του αθλητισμού και το οποίο ασχολείται με την Ε. Επίση θα υπάρχει και μια ανεπίσημη συνάντηση των Υπουργών Αθλητισμού που θα γίνει, καθώ επίση θα υπάρχουν και βασικοί πολίτε, σημαντικοί πολίτε που θα συμμετέχουν ε, για να τεθούν οι προτεραιότητε. Σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι να βελτιώσουμε την δημόσια υγεία και επίσης την κοινωνική συνοχή η οποία θα χρειαστεί. Σε αυτό το σημείο νομίζω πως το σπόρο, ο αθλητισμός μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο καθώς επίσης με την υπό την Βελγική Προεδρία υπήρξε ένα σιτό συντονισμό ο οποίο έχει γίνει και τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτό προσπάθησαν αυτή τη στιγμή να αναπτύξουν και ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο υιοθέτησε μια ε, πρόταση που είχε γίνει όσον αφορά την, υποστήριξη, την περαιτέρω υποστήριξη του αθλητισμού και νομίζω αυτό αποτελεί σταθμό για την ΕΕ αυτό που έχει γίνει μέχρι τούδε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. οι περισσότερες παρατηρήσεις ε, δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά υποσχόμενες διότι είπατε και αναφέρατε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία υπόληψη ενώπιον αυτού του προγράμματος για τον αθλητισμό δεν Κάναμε όμω τη δουλειά μα χθε. Διορίσαμε έναν εισηγητή για τα θέματα αθλητισμού που θα ασχοληθεί με την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφο μα Φίσερ. Γι' αυτό του δίνω αμέσω τον λόγο. Κύριε Φίσερ, παρακαλώ, και τον λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Και επιπλέον ίσως εξ ονόματος όλης της Επιτροπής μας ένας χαιρετισμό στον παλαιό συνάδελφο και πρόεδρο της Ουγγαρίας Παλ Σμιτ που είχε συνεργαστεί μαζί μα, Είναι ένα άτομο που πραγματικά είναι συνδεδεμένο με τον κόσμο του αθλητισμού και είμαι βέβαιο ότι θα υποστηρίξει τι προσπάθειε της Ουγγρική Προεδρίας και τη Ευρωβουλή για να αποκομίσουμε τα μέγιστα ωφέλη σε αυτό το θέμα. Τρει ερωτήσει θα ήθελα να σα διατυπώσω, συγκεκριμένε ερωτήσει. Πρώτα, υποθέτω ότι θα έχετε σίγουρα πληροφορίε ήδη για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Βασιλείου δηλαδή, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνιστώσας στον αθλητισμό. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια μια δεύτερη ερώτηση επίσης, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 για τον αθλητισμό. Σε τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Και εσείς αναφέρατε κάτι που μας ανησυχεί όλους πολύ. Είναι το πλαίσιο, το δημοσιονομικό σε σχέση με τον αθλητισμό. Εμείς θεωρούμε ότι ακριβώς τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αρμοδιότητες συγκεκριμένες και χειροπιαστές, με το άρθρο 165 της συνθήκης ε, της Λισαβόνας για τον αθλητισμό θα ήταν παράλογο να μην έχουμε ένα κονδύλιο στον προϋπολογισμό για τον αθλητισμό. Ξέρουμε ότι περνάμε μια περίοδο κρίσης αλλά αν η Ουγγρική Προεδρία μπορεί να κάνει κάτι για να ευνοήσει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον αθλητισμό καλό θα ήταν αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρούπελ, συνάδελφος, έχει τον λόγο, παρακαλώ. Uh, Έχουμε προβλήματα με τα μικρόφωνα, αλλά τώρα φαίνεται να λειτουργούν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αντιδράσω στις τοποθετήσεις που ακούσαμε γιατί τα όσα είπε η κυρία Βασιλείου λέει χθε το βράδυ. Πιθανότατα στη νέα μεσοπρόθεσμη αυτή η προοπτική το πρόγραμμα για τον αθλητισμό δεν εγγράφεται, δεν εντάσσεται και όλα τα άλλα προγράμματα που μας αφορούν περικόπτονται Μπορεί αυτό να φαίνεται πιεστικά πραγματιστικό, αλλά πολιτικά είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ανταποκρίνεται στη συνθήκη και στις νέες αρμοδιότητες που ζητούμε και έχουμε για τον αθλητισμό. Και οι νομοθέτες δημοσιονομικά είναι, εξακολουθούν και είναι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και βρίσκω ότι η κυρία Βασιλείου πρέπει να καταστήσει σαφέσα ότι δεν είναι δυνατόν τώρα το 2011 να γίνονται τέτοιες τοποθετήσεις διότι αντιβαίνουν την τάξη των πραγμάτων και θα ήθελα να ξέρω πώς η Ουγγρική Προεδρία θα αντιδράσει ή θα υπάρξει μια οξύ αντίδραση σε αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πάκολα, παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. αν ξεκινήσω με ένα φινοουγγρικό πνεύμα από αυτή την ομάδα εθνών, θα έλεγα σε σχέση με την Φινλανδία και το Υπουργείο ε, Παιδείας και Αθλητισμού για τις τοποθετήσεις που υπήρξαν. Αναφέρθηκε κάτι σε σχέση με το να κερδίζουμε μετάλλια λέει. Χαίρομαι πάρα πολύ ότι ο Ατήλας, ο Υπουργός δηλαδή, είναι ε, ο αρμόδιος για αυτό το θέμα, για αυτό το χαρτοφυλάκιο όχι ε, θα έλεγα σε ένα ε, ευρύτερο πλαίσιο αλλά μέσα στο δικό μας κύκλο έχουμε μεγάλες προσδοκίες από την, Φινλανδική, από την Ουγγρική με Προεδρία διότι γνωρίζουμε ότι οι δεσμεύσεις σας για τον αθλητισμό και για τι δεσμεύσει του Προέδρου του Παλ Σμιτ που βρισκόταν στην Ευρωβουλή παλαιότερα δεσμεύονται υπέρ του αθλητισμού. Σε μια περίοδο στην Ευρώπη που τα πράγματα δεν πάνε καλά οικονομικά χρειαζόμαστε επενδύσεις στον τομέα του αθλητισμού. Όταν επενδύει κανεί ένα ευρώ για τον αθλητισμό κερδίζει, εξοικονομεί δύο ευρώ όσον αφορά κοινωνικέ δράσει. Και ελπίζω ότι αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το μήνυμα, συγγνώμη, θα μπορέσει να περάσει και θα βρει αποδέκτες και θα ληφθεί υπόψη από άλλους ε, που διαμορφώνουν την πολιτική μας σήμερα. Φαίνεται ότι υπάρχει άγνοια σε σχέση με αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας προτρέψω, να σας ενθαρρύνω μια και έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ως Ουγγρική Προεδρία και έχετε και αυτό το άτυπο συμβούλιο για θέματα αθλητισμού από πλευρά των Υπουργών που θα διαξαχθεί στην Βουδαπέστη. Να το λάβετε υπόψη αυτό. Και οι προσδοκίες ε, όλων όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό και εμπλέκονται στο πεδίο είναι πολύ υψηλέ. Ε, ε, δίνεται προτεραιότητα. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα λοιπόν από πλευρά στον αθλητισμό. Είναι σημαντικό αυτό. Οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη πλευρά και από την Ευρωβουλή έχουμε μια νομική βάση αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα πλέον. Και θεωρώ ότι Κάνετε κάθε προσπάθεια, ό,τι περνάει από το χέρι σας. Θέλω να σας ενθαρρύνω λοιπόν. Τώρα που είναι η ώρα πρέπει να χτυπήσουμε το σίδερο για να κολλήσει. Και τώρα πρέπει να δραχθούμε τη ευκαιρία και να πιάσουμε δουλειά, να ανασκουμποθούμε, να ανασκουμποθούμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Συνάδελφος Μπόρις παρακαλώ. Ja również chciałem podziękować bardzo za to optymistyczne przedstawienie. Ευχαριστώ. Πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι παρακαλώ. Μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα, νομίζω πω η Κομισιόν είναι πάρα πολύ δραστήριο όσον αφορά τον αθλητισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τι βέλτιστε μεθόδου. Μερικά κράτη-μέλη και ιδιαίτερα η Ουγγαρία θα θέλανε να υπάρχει ένα πρόγραμμα πλαίσιο για τον αθλητισμό ούτως ώστε να γίνει μια επίσημη πολιτική της ΕΕ και να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Εξού και το ερώτημα κύριε Υπουργέ και θα θέλαμε να ξέρουμε σε όλες τις εργασίες οι οποίες θα γίνονται όσον αφορά τα πλαίσια χρηματοδότησης θα πρέπει για το 2014 θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι σωστέ πρακτικέ και νομίζω πω η νομική βάση μα επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο σα προτείνω να συνεχίσετε τι δραστηριότητε τι οποίε αναπτύσσετε και εμεί έχουμε μεγάλε ελπίδε από την Προεδρία σα, την Ουγγρική δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ήταν πολύ σαφής η ανασκόπηση της, ε, των προθέσεων της Ουγγρικής Προεδρίας. Θα ήθελα ε, ένα σχόλιο για τον αθλητισμό για την τρίτη ηλικία. Είναι ένα θέμα που δεν συζητήσετε ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα θα έχει ωφέλη από κοινωνική ε, άποψη και άποψη υγεία. Θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο τι προτίθεστε να κάνετε στον τομέα αυτό. Εκέσ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ, εάν υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορούμε να αποκαλέσουμε ευρωπαϊκό, τότε είναι το θέμα του αθλητισμού. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το μοιραζόμαστε όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρώπη, αλλά θα ήταν μεγάλο λάθος εάν δεν ε, θεωρούσαμε το πρόγραμμα του αθλητισμού ως αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω προς ε, την ε, Επιτροπή μας να ε, κάνει ό,τι μπορεί να διαθέσει όλα τα μέσα έτσι ώστε να θεσπιστεί και να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα στον αθλητισμό ως μέρος της στρατηγικής ε, Ευρώπης 2020. Ο, ο Υπουργός Τσένε προσκλήθηκε πρόσφατα στην Ρουμανία στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου Οράντα. Και αυτή είναι μια ένδειξη του πώς μπορεί να φέρει ο αθλητισμός κοντά τα κράτη και τα έθνη, διότι ο αθλητισμός είναι μια κοινή γλώσσα ανάμεσα σε όλα τα έθνη και όλα τα ε, και όλες τις χώρες. Μας φέρνει, κοντά. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω κλείνοντας είναι να, ε, να δώσουμε έμφαση στη νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δυσκολεύεται να μεταδώσει αυτό το πρόγραμμα στους πολίτες και αυτό είναι ένα συνεχές πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και ε, σε τελευταία ανάλυση ε, μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να απευθυνθούμε στους νέους. Άρα είναι μια προστιθέμενη αξία αυτό το πρόγραμμα σε θέματα αθλητισμού και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα με άλλα λόγια. Ποιες είναι οι πιθανότητες κύριε Υπουργέ αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί και τι μπορούμε να κάνουμε κυρία Πακ για να ε, ενταχθεί αυτό το πρόγραμμα στη στρατηγική 2020. Um, Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τα σχόλια του Υπουργού. Ε, και χαίρομαι που τα έχετε θέσει πολύ ψηλά ε, στις προτεραιότητες σας. Έχουμε αυξημένε προσδικίες για τα θέματα αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα και θα πρέπει να υπάρχει κονδύλι του προπολογισμού που να χρησιμοποιηθεί. Αλλά πρέπει να εντοπίσουμε πίσουμε στο χρόνο που έχουμε μέχρι το 2014 ακριβώς πού μπορεί να προσθέσει αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού μπορούν να έχουμε αποτελέσματα επιτόπου διότι ανησυχώ ότι μπορεί να πάρουμε τα χρήματα και, ε, ε, και η ερώτηση είναι πώς θα διασφαλίσετε ότι ε, θα δώσετε έμφαση και σε βασικά αθλήματα, όχι μόνο σε αθλητισμό ελίτ για, να συμμετέχουν και αυτοί πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ακουστούν και οι φωνές των, ε, των βασικών αθλημάτων. Ο, ο τελευταίος που θα παρέμβει ο κύριος Μικάρσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Υπουργέ. Αληθεύει Υπουργέ ότι η Ουγγρική Προεδρία πρόκειται να αναλάβει ειδική δράση, υπογραμμίζω το ειδική δράση στις δραστηριότητες σε σχέση με χώρες που βρίσκονται στο πρόγραμμα της Ανατολικής Γειτονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ, Τζένες, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. θα προσπαθήσω χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο χρόνο να απαντήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Πρώτα και κύρια, όσον αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της 18ης Ιανουαρίου που καλοχαιρετίστηκε όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό είναι ο τίτλος ε, με τους Ισπανούς και ε, Βέλγους ε, όσον αφορά τις προηγούμενες προεδρίες ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτής της ανακοίνωσης για αυτό το θέμα. Είναι η πρώτη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναλαμβάνεται μετά την έναρξη σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Και έχουμε φόρτο, έχουμε δουλειά που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα εργασίας και από κοινού τα κράτη-μέλη αυτό στοχεύουμε να κάνουμε σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτό ικανοποιεί ως απάντηση βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο λόγο για αυτό το θέμα αν επιθυμείτε. Ουσιαστικά θεωρώ ότι με βάση αυτή την ανακοίνωση μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την πραγματική δουλειά. Και τώρα δεύτερη ερώτηση. Πώς μπορεί ο αθλητισμός να συνεισφέρει σε σχέση με την επίτευξη ευόδοση της στρατηγικής για το 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό, μεγάλο δυναμικό σε αυτό το πεδίο. Και αυτό επειδή είναι και εξειδικευμένο ο αθλητισμός ως ζήτημα, αλλά είναι και οριζόντιο θέμα, εγκάρσιο θέμα για την επίτευξη διάφορων στόχων. Την καταπολέμηση, για παράδειγμα, του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την ένταξη την κοινωνική μειονεκτικών ομάδων κοινωνικά και να ε, προωθηθεί η κινητικότητα, η κινητικότητα, η απασχόληση, να βελτιωθεί η δημόσια υγεία. Επίσης εξάλλου μπορεί να μειωθεί ο αριθμός, ε, αν καλλιεργήσουμε τον αθλητισμό, ο αριθμό των ημερών κατά τον οποίο ασθενούν οι πολίτε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μιλήσουμε γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα πρόγραμμα πλαίσιο για τον αθλητισμό και γιατί πρέπει να βρούμε τα επαρκή κεφάλαια, τα κονδύλια για την χρηματοδότηση του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων των αθλητικών. Κάθε ευρώ στην ε, Ουγγαρία, λέμε κάθε ε, φλωρίνη που δαπανούμε για τον αθλητισμό, έχει ε, μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά και κέρδος για την κοινωνική πολιτική. Και αυτό πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στην πρώτη γραμμή της δράσης μας. Μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν σίγουρα ωφέλη, θα υπάρξουν κέρδη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ο αθλητισμός ως ε, μόνο αθλητισμός και δραστηριότητες σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο ή ανώτατο επίπεδο, δηλαδή των ε, ε, καλύτερων επιδόσεων. Μπορεί να υπάρχει και ευρύτερη ευρύτερο πεδίο για τον αθλητισμό, όπως για παράδειγμα για την τρίτη ηλικία, μπορεί να συνεισφέρει συνολικά ο αθλητισμός υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της Ευρώπης. Επόμενο θέμα η χρηματοδότηση από πλευράς προϋπολογισμού, τα δημοσιονομικά και τα κονδύλια. Έτη διαπραγματεύσεων προηγήθηκαν την έγκριση ενός προγράμματος πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει φυσικά να υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο βήμα, κοινή απόφαση που θα επιτυγχάνεται από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό ακριβώς που κάνω τώρα, αν θέλετε, είναι ασκώ πίεση, κάνω έργο λομπιίστα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ζητώ να υπάρξει η υποστήριξή σας, γιατί αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο είναι σημαντικό και πρέπει να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι αλλά και να κάνουμε και άλλους, να πείσουμε και άλλους ότι είναι κάτι παραπάνω ο αθλητισμός ως ευρύτερο συνολικό θέμα από ότι οι παγκόσμιες επιδόσεις, τα ρεκόρ και ε, ε, το κυνήγι των μεταλλίων. Δεν είναι το θέμα αν μπορεί κάποιος να κολυμπήσει ταχύτερα από κάποιον άλλο, αλλά είναι η δραστηριότητα η ίδια. Είναι λοιπόν ε, είναι κάτι το οποίο είναι διεθνές και όλοι το κατανοούμε αυτό. Για τους περισσότερους αθλητισμός όμως είναι τα είδωλα. Η, θα έλεγα ο εμβληματικός χαρακτήρας των καλύτερων αθλητών που λατρεύει ο κόσμος. Υπάρχει αυτό το ευρύτερο πλαίσιο λοιπόν όπως προανέφερα και ένα από τα θέματα αφορούσε τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των αθλητικών αυτών προγραμμάτων και δράσεων και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον αθλητισμό ε, συνολικά για τον λαό, για τον απλό κόσμο και όχι μόνο για τους καλύτερους αθλητές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αυτή τη διαφοροποίηση ώστε οι πολίτες, οι απλοί πολίτες να υποφερούνται στο μέγιστο. Στόχος μας πρέπει να είναι οι αθλητικές δραστηριότητες να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Χρειαζόμαστε τα αθλητικά είδωλα γι' αυτό. Χρειαζόμαστε τα πρότυπα, τα υποδείγματα. Χρειαζόμαστε τους ε, ρέκορντ με τους ε, αθλητές που είναι οι καλύτεροι παγκόσμια και για τους οποίους είναι περήφανες οι χώρες τους και είναι η περηφάνεια του, των πολιτών ώστε τα παιδιά με την υποστήριξη των γονιών και της οικογένειάς τους να αρχίσουν να αθλούνται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δεν κάνει διαφορά αν θα είναι επιτυχής στο παγκόσμιο επίπεδο ή απλώς αν θα ενασχολούνται με τον αθλητισμό και θα αγαπούν τα αθλήματα. Η Επίτροπος Βασιλείου έχει δεσμευθεί ιδιαίτερα και καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες. Πρέπει να δούμε όμως η κυρία Πάκος πρόεδρος αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, έχει συγκεκριμένους στόχους και στοχοθετημένα δρά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ακόμα. Και ήταν πολύ ευγενικό και καλό αυτό που ακούστηκε ότι δηλαδή υπάρχει πρόκληση που διατυπώνεται από πλευρά των μελών της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής ότι δεν έγιναν αρκετά όσον αφορά τον αθλητισμό και πρέπει να δοθεί μάχη για το πρόγραμμα αυτό μέχρι το 2013. Και από το 2014 εφ' εξής, μεταξύ 2014 και 2020 χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα πλαίσιο για τον αθλητισμό και πρέπει να βρούμε για αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο για τον αθλητισμό ποιο θα είναι ο τρόπο που θα επωφελήσει με τον καλύτερο τρόπο τα 27 κράτη-μέλη και πώ αυτά θα αποκομίσουν το μέγιστο κέρδο. Μέσα στην κάθε χώρα μας την ίδια θα πρέπει να εντάξουμε τον αθλητισμό και τις ε, αθλητικές δραστηριότητες ε, στη ζωή των χωρών μας για τον προϋπολογισμό του της, ε, για την νεότητα και τον αθλητισμό που άκουσα ότι περικόπτεν, υπάρχουν περικοπές ε, αυτό με θλίβει, αυτά συνδέονται αλληλοσυνδέονται, γι' αυτό έχουμε κοινέ αρμοδιότητες ε, όσον αφορά τις δικές μας δραστηριότητες και τους αρμόδιους στην, για αυτά τα θέματα στην Ουγγαρία. Είμαστε οι τέσσερις που εμπλεκόμαστε και που πρέπει να δούμε ότι ως ομάδα θα αντιμετωπίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο αυτά τα θέματα. Πρέπει να δούμε και τον αθλητισμό ως καθοριστικό παράγοντα και για την υγεία. Και τα κονδύλια που πρέπει λοιπόν να δαπανώνται πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοίχηση και με τα ωφέλη για την δημόσια υγεία το να σημαίνει ότι όταν δαπανούμε κάποια κονδύλια για τον αθλητισμό πρέπει να σφίγγουμε το ζωνάρι αλλού, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια αυτό πρέπει να μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα, αθλητισμός για την τρίτη ηλικία. Αυτό που μπορώ μόνο να πω είναι ότι η Ουγγρική Προεδρία θέλει να επικεντρωθεί στη, στον αθλητισμό για την τρίτη ηλικία. Και εγώ είμαι, μπορώ να πω πλέον, έχω πάρει κάποια χρόνια και σε, επίπεδο, σε τέτοιο επίπεδο θα μπορούσα πλέον να συμμετάσχω. Ακούσατε όλοι για το πρωτάθλημα και, τον, και την εμπλοκή των πρωταθλητών. Είδα ότι υπάρχουν και πολίτες άτομα της τρίτης ηλικίας σε, αγωνισμούς, σε διαγωνισμούς κολύμβησης, σε, στην κολύμβηση και είδα πολίτες που έμαθαν μόνο πριν από κάποια χρόνια και είναι της τρίτης ηλικία άτομα και έμαθαν να κολυμπούν. Και αθλούνται όμως, συναγωνίζονται, ανταγωνίζονται άλλους και συμμετέχουν σε τέτοιους κολυμπητικούς αγώνες, αγώνες κολύμβησης σε άλλα κράτη-μέλη. Αν μπορέσουμε κάποιες χιλιάδες άτομα και τις οικογένειές τους να τις προσελκύσουμε με αυτόν τον τρόπο, να τις κινητοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε κάποιες χιλιάδες άτομα, ήδη θα έχουμε πετύχει πάμπολα. Όσο περισσότερα άτομα κινητοποιούμε με την ε, προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω των αθλητικών δραστηριοτήτων, τόσο μεγαλύτερη απήχηση θα έχουμε στους πολίτες μας και τόσο περισσότερο θα είναι το όφελος. Μπορούμε και σε σχέση και με τις γυναίκες ε, να πούμε τα ίδια. Και ένας άλλος τομέας που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό και με άλλα θέματα είναι ακριβώς αυτό. Ο αθλητισμός πρέπει να είναι κάτι που θα είναι προσπελάσιμο και ανοιχτό για συμμετοχή όλων. Όλοι πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το φύλλο ή την ηλικία τους. Και ελπίζουμε λοιπόν τούτων λεχθέντων ότι η Ουγγαρία θα καταφέρει να φτάσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε το 30-32% των ε, Ούγγρων να ασχολούνται τακτικά και ε, πιο συχνά με τις ε, αθλητικές δραστηριότητες. Αυτό είναι εκείνο που πρέπει να πούμε. Για μένα ως αθλητή η καθημερινή ενασχόληση με τον αθλητισμό, η εβδομαδιαία ενασχόληση μια μισή ώρα την ημέρα τρεις φορές την εβδομάδα είναι σημαντική υπόθεση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η προσέγγιση και η νοοτροπία των πολιτών. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που επιθυμούμε να επιτύχουμε και αυτό που είναι εφικτό και μπορεί να γίνει και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη χρηματοδότηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια και ήμουν Ολυμπιακός ε, ε, πρωταθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχω το σθένος και στοχοθετώ ε, πράγματα ώστε να μπορώ να δώσω τη μάχη αποτελεσματικά. Βλέποντας ότι είναι σημαντικός ο αθλητισμός και το πρόγραμμα πλαίσιο για τον αθλητισμό μέσα ή σε αυτή την συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και εκτός αυτού έχω πιστεί ότι αξίζει τον κόπο να δώσει κανείς τη μάχη υπέρ αυτού. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη αλλά έχω την υποστήριξη και χαίρομαι γι' αυτό των οπαδών και στην Ουγγαρία θα έχω την δική σας υποστήριξη και με τη δική σας λοιπόν υποστήριξη και σύνδρομη θα είμαι σε θέση να, να... να αγωνιστώ, να δώσω μάχη ώστε να προχωρήσει ο αθλητισμός και να διασφαλίσουμε τα κονδύλια που είναι αναγκαία. Νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες από τις ερωτήσεις παρεμβάσεις. Ελπίζω ότι κατάφερα να απαντήσω τις πιο σημαντικές από ε, τις ανησυχίες σας. Αν έχετε κάποιο άλλο θέμα είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ πολύ. Προσέξτε, θα ήθελα μόνο να παρατηρήσω κάτι. Είναι μια ε, κάτι ανεκδοτολογικό αυτό όταν έχουμε για πρώτη φορά τα θέματα αθλητισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας και σε αυτό το επίπεδο κιόλα αμφισβητούνται από κάποιου ε, αυτά τα πράγματα. Όχι όμω από εμά. Όταν η ίδια η Επίτροπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν υπόψη το ψαλίδι και να αρχίσουν να περικόπτουν κονδύλια, δεν θα γίνει τίποτα στο τέλο. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Όλα θα πάνε του κάκου. Δεν χρειάζεται να απευθύνεται σε εμά έκκληση, κύριε Υπουργέ, να δώσουμε εμεί κονδύλια. Δεν είμαστε εμεί που διαθέτουμε τα κονδύλια. Εσεί, το Συμβούλιο, δίνετε τα κονδύλια. Πρέπει να μιλήσετε με του ομολόγου σα, τον Ολλανδό, τον Γάλλο, τον Γερμανό συνάδελφό σα και το δικό σας Υπουργό Οικονομικών. Οι Υπουργοί Οικονομικών λοιπόν πρέπει να πιστούν. Ο αγώνας πρέπει να ξεκινήσει τώρα αμέσω ώστε να μην γίνει πραγματικότητα η απειλή της ψαλίδας και των περικοπών. Δεν γίνεται να αληθεύει ότι δεν θα υπάρξει πρόγραμμα, λέει, όπως ακούγεται από κάποιες φήμες. Φίλοι, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και οι κυρίες και κύριοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ να διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα στους υπεύθυνου της Επιτροπής. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το ίδιο επιθυμεί όπως και εμείς, γιατί διαφορετικά δεν θα έκανε την ανακοίνωσή της, θα μπορούσε τότε να μην έκανε τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε δεκάρικους λόγους, αυτή είναι ανώφελη. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είμαστε εδώ και στοχοθετημένα εσείς πλειοψηφικά ε, μπορεί κανεί να τα λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εσεί είσαστε όμω οι αρμόδιοι από το Συμβούλιο που διασφαλίσετε τα κονδύλια. Και η κυρία Επίτροπο πρέπει να έχει στένο και να προσπαθεί να πετύχει αυτά που επιθυμούμε και εμεί να πετύχουμε. Τότε ίσω καταφέρουμε κάτι. Αν όλοι λένε δεν θα βρεθεί χρηματοδότηση, τότε γιατί κάνουμε λόγο και γιατί αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, εσεί θα δώσετε τη μάχη και θα υπάρξουν τα κονδύλια. Η κυρία Ρώσα Χόφμαν στη συνέχεια. Η κυρία Υπουργό, παρακαλώ. die Staatsministerin. Aha, ja. You understand that? Yes. Λοιπόν, σα καλοχαιρετίζουμε με τους συναδέλφους μας και από πλευράς εισηγητού που είχε ε, ασχοληθεί με το θέμα για την κινητικότητα μπορούμε να το η κινητικότητα των νέων. Και για, μέσα στο πλαίσιο της κινητικότητας ε, της ε, νεολαίας και της νεότητας ε, μπορεί να δει κανεί όλα τα προγράμματα που χρειαζόμαστε, όλα τα προγράμματα παιδείας και εκπαίδευσης, το πρόγραμμα για την νεότητα, για τους νέους, το πρόγραμμα για τον αθλητισμό που ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, θα αποκτήσει σάρκα και οστά. Και γι' αυτό πιστεύουμε και λέμε ότι υπάρχει κάθε συμφέρον και ενδιαφέρον τώρα στη δική σας Ουγγρική Προεδρία να θέσετε τη σωστή, να χαράξετε τη σωστή πορεία ώστε έγκαιρα να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα προγράμματα αυτά για την παιδί την εκπαίδευση. Έχετε τον λόγο, 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας και ακριβώς όπως με τον συνάδελφό σας θα τεθούν ερωτήσεις στη συνέχεια. Παρακαλώ έχετε τον λόγο λοιπόν κυρία Υπουργέ. Μια στιγμή. Εσείς που βρίσκεστε εκεί πίσω, προσπαθήστε να βρείτε κάποια θέση να καθίσετε. Υπάρχουν κάποια κενά έδρανα. Μπορείτε να βρείτε να καθίσετε. Λοιπόν. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Τέλος πάντων, εντάξει. Ήθελα να σας βοηθήσω. Είστε τον λόγο κύριε Υπουργέ. Αντιμαμέλη, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα ως Υπουργός Αρμόδιος για θέματα παιδείας ε, να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας για να δώσω την αναφορά σχετικά με τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας στο θέμα της παιδείας. Χαίρομαι να αναφέρω ότι σύμφωνα με την γνώμη των εμπειρογνωμόνων μας είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την Προεδρία. Το είχε αναφέρει και ο κύριος Μπαρόσο στη Βουδαπέστη στις αρχές Ιανουαρίου και έχουμε ένα έγγραφο του προγράμματος, παρόλο που δεν επισέρχεται σε λεπτομέρειες θέματα παιδείας, στη σελίδα 49 μπορείτε να δείτε μία περίληψη των θεμάτων που άπτονται της παιδείας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, τον περασμένο ε, Ιούλιο θεώρησαν την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως σημαντικό μέρος του μέλλοντος της Ευρώπης. Συνεπώς, ε, στην θητεία αυτή θα προσδώσουμε μεγάλη σημασία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και προσωπικά έχω δεσμευτεί στο θέμα της παιδείας, διότι έχω αφιερώσει την σταδιοδρομία μου ως εκπαιδευτικός, μετά ως μέλος της Βουλής, έχω ασχοληθεί με θέματα παιδείας, έχω προσωπική εμπειρία λοιπόν σε θέματα, στο θέμα της αρμοδιότητάς μου και επίσης αυτό που συμβαίνει σήμερα στα σχολεία θα διαμορφώσει την κοινωνία του μέλλοντος. Ως αυτού του η παιδεία είναι πρώτη τη σημασία για μένα και κατανοώ ότι η εκπαίδευση δεν είναι θέμα ε, λεφτών. Βέβαια, μια καλή παιδεία μπορεί να στοιχίζει πολλά, αλλά χρειάζονται και καλά προγράμματα. Άρα η δαπανερή παιδεία είναι καλή μόνο αν υπάρχουν καλά προγράμματα με καλά αποτελέσματα και καλά ορισμένους στόχους. Είμαι μέλος, είμαι μέλος της Βουλής εδώ και πέντε χρόνια, γι' αυτό καταλαβαίνω ακριβώς πώς λειτουργούν τα κοινοβούλια και χαίρομαι που σας γνωρίζω και θέλω να σας διαβεβαιώσω σε αυτό το σημείο ότι κατά την θητεία της Ουγγρικής ε, Προεδρίας και στη συνέχεια θα είμαι στη διάθεσή σας βέβαια. Επίσης θα ήθελα να σας καλέσω σε όλα τα γεγονότα, όλα τα συνέδρια που θα διοργανωθούν στα πλαίσια αυτού του εξαμήνου στην Βουδαπέστη, στον Κέντολο και θα προτείνουμε πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, συναρπαστικά προγράμματα που μπορεί να μην ε, μεταμορφώσουν βέβαια τον κόσμο εν μία νυχτή, αλλά θα ε, δώσουμε συνέχεια σε θέματα ε, που τονίζουν το ρόλο της παιδείας. Αυτό το εξάμεινο είναι μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι και το πρώτο εξάμεινο. Ο... Ξεκινάει λοιπόν ε, στις 12 Ιανουαρίου ε, δημοσιεύθηκε μια έκθεση και αναλάβαμε λοιπόν το καθήκον να ε, διαχειριστούμε λοιπόν τις εργασίες του πρώτου εξαμήνου. Για, στην προετοιμασία μου για τη σημερινή συνεδρίαση διάβασα την ε, ετήσια ε, έκθεση της μεγένθησης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες οι δημοσιονομικές από την Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω ότι σύμφωνα με αυτή την έρευνα οι προτεραιότητες ε, δίδονται σε τομείς που απτούνται του Τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Γι' αυτό τονίζονται οι τομεί τη έρευνα, τη ε, εκπαίδευση ε, και τη ενεργειακή πολιτική. Η έρευνα μεγέθυνσης είναι μια σωστή αναπαράσταση των στρατηγικών στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική 2020. Και θα έλεγα ότι δίνουν μια ανατροφοδότηση και μια επιβεβαίωση της στρατηγικής, των, των στόχων στρατηγικής 2020, ε, όπου θα ήθελε να συνεισφέρει και η Ουγγαρία με αποφασιστικό τρόπο. Άρα οι περιεκτικές προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας οι περισσότερες, ε, τις οπερατήρες ε, τις ε, συνεχίζουμε από τις προηγούμενες τις προεδρίες, Ισπανικής και Βελγικής προεδριών και η υλοποίηση της στρατηγικής 2020 είναι παραγοντές που καθορίζουν το πρόγραμμά μας και θα συνεισφέρουν σε μια ισχυρότερη, μεγαλύτερη, πιο ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο δυνατή. Θα ήθελα να τονίσω αυτό, ιδιαίτερα στο θέμα της παιδείας. Πώς μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα σε αυτούς τους στόχους, μεγαλύτερη, πιο περιεκτική, πιο ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, ισχυροποιώντας τη στρατηγική 2020 αφενός, ενισχύοντας την, όπου η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να έχουν κομβικό ρόλο. Οι το όχι της στρατηγικής στο θέμα της εκπαίδευσης, ε, τους οποίους πρέπει να υλοποιήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας για αυτό το εξάμεινο. Για μια πιο περιεκτική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, η Ουγγρική Προεδρία θέλει να προωθήσει ε, την ε, ε, καλλιέργεια των αξιών της διαφορετικότητας. Έχουμε δει την μελέτη εκ νέου των δημογραφικών προβλημάτων και των πιο επιγόντων προβλημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού, πολέμηση της ένδυας ανάμεσα στα παιδιά και επίσης δημιουργία ενός πλαισίου για τη στρατηγική συμπερίληψης και ένταξης των Ρωμά. Ε, οι κυρίαρχες πτυχές ε, του πλαισίου ε, εκπαίδευση είναι η ενίσχυση της κοινωνικής πτυχής. Θέλουμε να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους για την διαβίου μάθηση και θέλουμε να τονίσουμε τα πρώιμα στάδια της εκπαίδευση για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη τώρα. Μπορούμε να δούμε αν η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να φέρουν ωφέλη που θα έχουν άμεσο και έμεσο αντίκτυπο στην οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη έτσι ώστε να κάνουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο σταθερή, πιο ανταγωνιστική στην διεθνή αρένα. Ε, τώρα θα ήθελα να επισέλθω σε κάποιες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της ε, Ουγγρικής Προεδρίας. Όπως είπα, η σημαντικότερη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση της στρατηγικής 2020 και η έγκριση ε, των θέσεων του Συμβουλίου. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ε, βελτίωση της ποιότητας της πρωτοβαθμιάς παιδείας και αύξηση της συμμετοχής. Ε, οργανώνουμε συνέδριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το τρίτο είναι η αποτροπή ε, της εγκατάλειψης ε, του σχολείου σε πρώιμα στάδια και θα θέλαμε και εκεί να εγκριθεί μια θέση του Συμβουλίου. Κινητικότητα πρέπει να προωθηθεί και ε, θέλουμε να εγκριθούν ε, συστάσεις του Συμβουλίου σε αυτή τη θητεία της Προεδρίας. Θα ήθελα να δώσω και κάποια άλλα θέματα που, στα οποία θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην Προεδρία αυτή, στο θέμα της παιδείας. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση. Αυτό είναι καταφανές το γεγονός ότι περίπου 50% των μαθητών και φοιτητών ε, φτάνουν σε επίπεδα λυκείου και στην ηλικία των 25 34 από τους τρεις μόνο ο ένας είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου δεν είναι θετικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τα 60 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης που χρειαζόμαστε μέχρι το 2020 θα απαιτούν υψηλότερα επίπεδα παιδείας και επίσης υποθέτουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ε, κατά 12 εκατομμύρια θέσεις λιγότερες. Ε, άρα υψηλότερα προσόντα είναι κάτι το οποίο θέλουμε να τονίσουμε στην Προεδρία μας. Και αυτό είναι αλληλένδετο με μια άλλη προτεραιότητα, δηλαδή τα, ε, η εκπαίδευση στα πρώτα επίπεδα. Από εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής πλευράς έχει αποδειχθεί ότι παιδιά τα οποία δεν εκπαιδεύτηκαν στα πρώιμα στάδια της παιδείας χάνουν ε, τις ε, ε, πιθανότητες τους να έχουν προσόντα που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βρουν θέσεις απασχόλησης και να γίνουν χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία. Άρα τα, η πρωτοβάθμια παιδεία είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο τονίζουμε. Η Επιτροπή θα ήθελε να θα μεταδώσει μια ανακοίνωση σε αρχές Φεβρουαρίου και θα οργανωθεί ένα συνέδριο με βάση αυτή την ανακοίνωση και θα θέλουμε να δούμε την έγκριση των στάσεων του Συμβουλίου μέχρι το Μάιο του 2011. Για να μειώσουμε το βαθμό εγκατάλειψης ε, αυτό είναι ένα άλλο αλληλένδετο σημείο και μια προτεραιότητα της Ουγγρικής ε, Προεδρίας και επίσης σχετίζεται με τη στρατηγική για την συμπερίληψη των Ρωμά. Στην ε, Βουδαπέστη ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Η νέοι εν κινήσει, κινητικότητα των νέων» που θα ακολουθήσει και σε άλλες πρωτεύουσες έχουμε δεσμευθεί στους στόχους και σε αποτέλεσματα για να αυξήσουμε τον αριθμό των μαθητών και φοιτητών που συμμετέχουν ε, σε αυτό το πρόγραμμα στο 20%. Δεν είναι καινούργια προτεραιότητα, είναι μια παράδοση που ξεκίνησε εδώ και αιώνες και ε, αυτό βοηθά στο άνοιγμα της Ευρώπης και στη βελτίωση των πιθανότητων απασχόλησης των νέων μας. Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ στην ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Το 2011 είναι το έτος εθελούσιων δραστηριοτήτων για την ενεργό πολιτότητα. Και στις 28 και 29 Μαρτίου οργανώνουμε ένα συνέδριο ε, με μια πολύ συναρπαστική ημερήσια διάταξη. Θα συζητήσουμε τις δεξιότητες, αρμοδιότητες και γνώσεις που απαιτούνται να έχουν οι νέοι έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατία, να συνεισφέρουν στις ε, κοινωνίες με υπεύθυνο τρόπο. Θα λάβουμε υπόψη επίσης τους παράγοντες που θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη στα σχολεία για να ενισχύσουν αυτό το δυναμικό. Θα συζητήσουμε επίσης ένα αρνητικό φαινόμενο το οποίο είναι η βία στα σχολεία και η επιθετικότητα και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη βία στα σχολεία. Και ε, τέλος ε, θα ήθελα να συζητήσω ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο προτείνουμε να θέσουμε ε, στην ατζέντα, δηλαδή την υποστήριξη των πρικισμένων παιδιών. Ε, τον Απρίλιο θα, είναι ε, θα γίνει ένα συνέδριο που θέλουμε να οργανώσουμε ε, για ανταλλαγή απόψεων στο θέμα αυτό. Γνωρίζοντας την ιστορία της Ευρώπης, συμφωνούμε όλοι ότι τα ταλέντα, τα πρικισμένα άτομα μπορούν να προωθήσουν την πρόοδο στον κόσμο και μπορούν επίσης να βοηθήσουν άλλους στο να κερδίσουν γνώσεις. Και η υποστήριξη των ταλέντων συσχετίζεται σε σχέση με το σύνολο της κοινωνίας. Συνολικά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάθε παιδί, κάθε άτομο έχει κάποια ταλέντα. Είναι, έχει, έχει πρικιστεί με κάποια ταλέντα και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ της Ευρώπης, κυρίως από πλευράς εκείνων των νέων που έχουν εξαιρετικά τέτοια τάλαντα. Θα πρέπει αυτοί να υποστηριχθούν, να τους συνδράμουμε. Αυτή θα είναι η πηγή των καινοτόμων μέτρων και πρωτοβουλίων που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα επωφελήσουν συνολικά την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό θα θέλαμε να υποβάλουμε συστάσεις για μια Ευρωπαϊκή ημέρα πρικισμένων ανθρώπων, ε, ταραντούχων θέλαμε να έχουμε την υποστήριξή σας να γίνει αυτή η πρωτοβουλία πραγματικότητα, να αποκτήσει σάρκα και οστά και να κινητοποιηθούμε υπέρ αυτής. 25η Μαρτίου είναι η ημερομηνία, η μέρα γέννησης που γιορτάζουμε τα γενέθλια, τη γέννηση του Μπέλα Μπάτοκ, του μεγάλου Ούγγρου συνθέτη. Θέλουμε να, αυτή η μέρα να είναι η μέρα υπέρ των ταλαντούχων νέων στην Ευρώπη και άλλα θέματα που δεν θα συζητήσω τώρα εξειδικευμένα. Θα βρείτε πληροφορίες για αυτά όλα τα συναφή θέματα στα, στους φακέλους σας. Θα ήθελα όλους να σας προσκαλέσω αθρώα να συμμετάσχετε από πλευρά της Ευρωβουλής πολυάριθμοι να συμμετάσχετε και ελπίζουμε ότι σε αυτό το εξάμεινο θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ώστε να υποστηριχθεί η δραστηριότητα αυτή υπέρ της παιδείας εκπαίδευσης και των μέτρων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα σχολεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόφμαν. Τώρα έχουμε έξι συναδέλφους που ζήτησαν να παρέμβουν. Η κυρία Μπαντία Κουτσέτ παρακαλώ πρώτη. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για τις επεξηγήσεις σας και για το ότι ήρθατε σήμερα εδώ για να μας πληροφορήσετε για το τι σκέπτεστε να κάνετε ως Ουγγρική Προεδρία. Θεώρησα, ε, κατάλαβα αμέσα στο ευρύ φάσμα θεμάτων που εσείς ε, σχολιάσατε και θέσατε ότι βρίσκονται σε αυτό το φάσμα όλα τα θέματα που αφορούν την κατάτηση και την εκπαίδευση. Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα θέμα κυρίως για την επαγγελματική κατάρτιση, διότι ακριβώς εργαζόμαστε ε, για μια έκθεση για αυτό το θέμα, για την ευρωπαϊκή επαγγελματική κατάρτιση. Είπατε κάποια στιγμή, δεν είναι όλα, δηλαδή σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση δεν εξαρτώνται όλα από τα κονδύλια. Συμφωνώ μαζί σας επ' αυτού. Είναι όμως τα κονδύλια τα χρήματα πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Χωρί μεγαλύτερη χρηματοδότηση δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή ζούμε μεγάλε μεταβολέ στην κοινωνία μα. Έχουμε την οικονομική, δημοσιονομική κρίση, την ψηφιακή εποχή. Βρισκόμαστε μπροστά στη δυνατότητα η Ευρώπη πραγματικά να έχει ένα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει και να υπομειστεί στην παγκόσμια οικονομία ή δεν θα διαδραματίσει κανένα ρόλο αν δεν τα καταφέρει. Όλα περνάνε από μένα από την καλύτερη παιδεία, εκπαίδευση και κατάρτιση. Μέσα από αυτό υπάρχει ένα σημαντικό θέμα να δώσουμε μεγαλύτερο κύρο όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση σε όλα τα συναφή θέματα. Είπατε επίσης ότι έχουμε λίγους πτυχιούχους στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ πιθανότατα ή την Ιαπωνία. Αλλά επίσης μπορούμε να το πούμε και το βλέπουμε στα διαφορετικά κράτη-μέλη ότι υπάρχουν πολλοί πτυχιούχοι που δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενο που σπούδασαν. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση για το πώς εκπαιδεύουμε τους πολίτες μας και στις ανάγκες που έχει ίδια η αγορά και πρέπει να καλυφθούν. Είναι λοιπόν σημαντικό όταν προχωράμε σε αυτή την βελτίωση της κατάρτισης να έχουμε μια αντιστοίχηση και ένα συντονισμό με τις επιχειρήσεις να ακούμε πραγματικά πραγματικά τι χρειάζονται και υπάρχει και μια μάχη την οποία έχουμε μισοχάσει, μισοκερδίσει όσον αφορά την, ε, το θέμα αυτό. Είναι η γνώση των γλωσσών. Όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά επίσης και για τους καθηγητές που εκείνοι πρέπει να προωθήσουν αυτό το θέμα, να το προαγάγουν και να ε, κάνουν τους πολίτες να κινητοποιηθούν. Είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχετε μπροστά σας ως Προεδρία. <clears throat> Έχετε όλους τους υπουργούς βέβαια για την ε, παιδεία και εκπαίδευση που έχουν υποστεί περικοπές από την ψαλίδα <laughs> για τα κονδύλια. Θα ήθελα να ακούσω την δική σας άποψη, διότι νομίζω το κατάλαβα ότι δεσμεύεστε κατά όλων αυτών των πολιτικών περικοπών. Θα ήθελα να σας ακούσω να λέτε ότι η δέσμευση και η μάχη που θέλετε να δώσετε ακριβώς στις συνεδριάσεις ε, με τους ε, συναδέλφους σας ε, από τα διαφορετικά κράτη να δοθεί αυτή η μάχη ώστε η ψαλίδα να μην χτυπήσει την κατάρτιση και την εκπαίδευση. Θα έλεγα ότι είναι η μόνη από τις πολιτικές που θα γινόταν τεράστιο λάθος αν υπήρχαν περικοπές επ' αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για τις επεξηγήσεις σας. Και εγώ πιστεύω ότι σε σχέση με τις αρμοδιότητές σας, από ό,τι γνωρίζω, έχετε και το θέμα της έρευνας. Κάνετε λόγο για το τάλαντο και τους πρικισμένους ανθρώπους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως γνωρίζετε, Υπουργέ, το 2009 ήταν το έτος που αφιερώθηκε στη δημιουργικότητα και στην καινοτομία στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για παράδειγμα να αναπτύξουμε επίσης τις υποτροφίες Marie Curie, να τις αναπτύξουμε που επιπλέον είναι θέμα της Επιτροπής Πολιτισμού και εμείς έχουμε αρμοδιότητες όσον αφορά θέματα έρευνα σχετικά. Και εμένα πολλές φορές με ανησυχεί το ότι στην έρευνα οι ερευνητές μας στο τέλος τέλος πρέπει να μετακινούνται, να πηγαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε για να αποκτήσουν την αναγνώρισή τους. Έχουμε ε, τα βραβεία Νόμπελ που είναι μεν Αμερικανοί αλλά είναι ευρωπαϊκή ε, προέλευση οι περισσότεροι. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για αυτό το θέμα στην Ευρώπη και από πλευρά τη Ουγγρικής Προεδρίας για να προωθεί, να προωθηθεί η έρευνα στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Σα <clears throat> eh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εδώ να συγχαρώ πρώτα απ' όλα την Ουγγρική Προεδρία. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι ευρύτατο και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να πετύχετε να μεταμορφώσετε αυτό το πρόγραμμα και τις προτάσεις σας ε, και να αποκτήσει σάρκα και οστά στην πραγματικότητα χειροπιαστά. Με εξέπληξε ότι δίνεται τόση προσοχή στον, στα θέματα πολιτισμού, στην, στα θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, στον αθλητισμό και στα ζητήματα των Ρωμά, των Τσιγκάνων. Και για τους Ούγγρους που ίσως κάποιος θα έλεγε ότι θα ήθελα να το αποκρύψουν αυτό το θέμα, να το αποσιωπήσουν. Όχι, το έχετε εντάξει ως προτεραιότητα το θέμα των ε, Τσιγκάνων και θέλω και να ευχαριστήσω και γι' αυτό. Οι προτεραιότητες σας είναι προτεραιότητες και δικές μας επίσης σίγουρα για την Ευρωβουλή. Και κυρίως για μας ε, που είμαστε μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και εξετάζουμε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Νομίζω θέσατε το δάκτυλο επί του τύπου των ύλων και πραγματικά όπως προαναφέρθηκε ίσως θα χρειαζόταν να δοθεί μια μεγαλύτερη προώθηση στην επαγγελματική κατάρτιση και στην δυνατότητα επαγγελματικής ε, ε, αναγνώρισης μέσω πτυχίων, διπλωμάτων και μέσα από την διαδικασία της Κοπενχάγης και μια μεταρρύθμιση επίσης της ε, διαδικασίας στην ανώτατη εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μαρή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 Ευχαριστώ ε, Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Σχετικά με τη στρατηγική της Ευρώπης 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, προτείνει πέντε στόχους, κύριους στόχους, που θα πρέπει να επιτευχθούν από την Ένωση μέχρι το 2020. Δύο από αυτούς τους στόχους είναι στενά συνδεδεμένοι με τα προβλήματα τα οποία συζητάμε και εμείς σήμερα εδώ. Δηλαδή την μείωση των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια, μείωση θα πρέπει να είναι κατά 20 εκατομμύρια τουλάχιστον πολιτών και επίσης μείωση της αποχώρησης, της πρώιμης αποχώρησης από το σχολείο που πρέπει να κατέβει στο κάτω του 10% ένα στόχος που σχετίζεται ε, ε, επίσης κάτι άλλο, 40% θα πρέπει να έχουν το βάθμιο εκπαίδευση. Πού εκδηλώνεται περισσότερο, πού εκδηλώνονται αυτά τα προβλήματα τον πληθυσμό των Ρώμ, στους οποίους αναφερθήκατε. Και η ερώτησή μου είναι πώς εσείς διαβλέπετε στην πράξη αυτούς τους στόχους να εφαρμόζονται μέσα στους ΡΟΜ δηλαδή σε σχέση με την φτώχεια, την εγκατάλειψη από το σχολείο, διότι είναι σαφές ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή τι στόχους ή πώς βλέπετε τη σχέση ανάμεσά τους, πώς νομίζετε ότι θα πετύχουμε πράγματι να μειώσουμε την αποχώρηση από το σχολείο σε αριθμούς αφενός και ε, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ε, και βέβαια συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, τι μέτρα ή τι συγκεκριμένους στόχους έχετε μελετήσει σχετικά με το, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικής Εργασίας. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κάθε ε, επιτυχία. Uh, thank um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για αυτή την πολύ περιεκτική παρουσίαση. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ που δώσατε τις προτεραιότητες ε, στην νηπιακή εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντική αυτά τα χρόνια φυσικά και χαίρομαι που έχετε θέσει αυτή την προτεραιότητα. Ε, δεν έχω κάποια ερώτηση γι' αυτό, διότι έχετε, καλύψει, έχετε καλύψει ένα μεγάλο μέρος, αλλά θέλω να ρωτήσω ε, σχετικά με το θέμα των γλωσσών. Ε, αν είμαστε σοβαροί στο θέμα της κινητικότητας, είναι σημαντικό οι νέοι μας να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Και γνωρίζω σε, σε κάποια ε, κράτη-μέλη καλύτερα από άλλα, εμείς οι Βρετανοί ιδιαίτεροι δεν είμαστε καλοί στο να μαθαίνουμε γλώσσες. Είναι σοβαρό το ερώτημα, διότι δεν θα πετύχουμε την κοινικότητα, δεν θα υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Θέλω να δω τις απόψεις σας και να δω αν η Ουγγρική Προεδρία έχει οποιαδήποτε σχέδια προώθησης της εκμάθησης των γλωσσών. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμα. Τέκης Παλιατέλη καβέντα Μετά έτσι θα ολοκληρώσουμε. Τέκης παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, σας συγχαίρω για τα φιλόδοξα σχέδιά σας. Ο Ούγγρος και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που έχετε ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο. Πρώτη παρατήρηση. Σχετικά με την ε, ενσωμάτωση Ανατολής και Δύσης. Στο παραπέτασμα εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και εικονικά ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση της Ευρώπης. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παραμένουν πίσω σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής ε- Ευρώπης και αυτό οφείλεται κυρίως ε, στην ποιότητα και στο επίπεδο εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στην κοινότητα των ΡΟΜ είναι ένα τεράστιο εμπόδιο ε, στην ενοποίηση της Ανατολικής ε, και Δυτικής Ευρώπης σε μια Ενωμένη Ευρώπη. Εγώ βλέπω την εκπαίδευση ως ένα εργαλείο ενοποίησης και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο της εκπαίδευσης και τη, ε, η στρατηγική για τους ΡΟΜ είναι μια στρατηγική στην οποία θέλω να σας συγχαρώ, Σουγκρική Προεδρία, διότι ο μόνος τρόπος να ενσωματώσουμε την μειονότητα αυτών των ευπαθών ομάδων στην κοινωνία είναι μέσα από την εκπαίδευση. Το δεύτερο σχόλιο μου αφορά την, τις γλώσσες και τα θρησκευτικά. Μπορούμε να δούμε ότι οι Ρουμάνοι στην Σερβία οι Ουκρανοί στη Ρουμανία, υπάρχουν διακρίσεις ε, κατά των Ούγγρων στη Ρουμανία. Θα πρέπει... Αυτό είναι, ε, αυτό είναι γεγονός. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε δει εξελίξεις σε αυτό τον τομέα. Αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε ένα ουγγρικό πανεπιστήμιο για τα θρησκευτικά σχολεία, τα καθολικά ε, σχολεία, τα σχολεία της Εκκλησίας ε, τη χάνουν διακρίσεων στον τομέα της παιδείας. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό. Είναι θέμα δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Παλιατέλη, η εισηγήτριά μα για, ε, για την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Αυτό το θέμα θα το εξετάσουμε στη συνέχεια. Κυρία Παλιατέλη. Να ευχαριστήσω και την Υπουργό για την παρουσίαση, των ε, προτάσεων σχετικά με την Προεδρία στη διάρκεια τους, της Άνοιξης. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις, κυρία Υπουργέ. Ε, θεωρώντας ότι η παιδεία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ευρωπαϊκή συνοχή και όχι μόνο των μειονοτήτων όπως είναι η ρωμά αλλά και ανάμεσα στους λαούς όπως περιγράφηκαν πριν από λίγο από τον συνάδελφο. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να σκεφτείτε τη χρήση της ιστορίας, της γνώσης της ευρωπαϊκής ιστορίας ως ένα τέτοιο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και ένα δεύτερο ε, σύντομο ερώτημα. Έχουμε διαπιστωμένη μία τάση των ε, ευρωπαϊκών πανεπιστημίων να μειώνουν και τα κονδύλια και ε, ε, ε, που έχουν σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές. ποια πρωτοβουλία θα μπορούσατε να αναλάβετε στη διάρκεια της Προεδρίας σας προκειμένου να αποθαρρυνθεί μια τέτοια τάση που δυστυχώς κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην προοπτική της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε άλλες υπήρους. Ευχαριστώ πολύ. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Υπουργέ. Εντάχει, είμαστε όλοι πάρα πολύ ευαίσθητοι όλοι σε αυτά τα οποία είπατε όσον αφορά ε, παιδεία και ενσωμάτωση και ένταξη. Εγώ θα επιστιαστώ περισσότερο στους ΡΟΜ Ξέρετε, οι νότιες χώρες της Ευρώπης γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το θέμα. Οι Ρώμοι είναι Ευρωπαίοι όπως εσείς και εγώ. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι είναι νομάδες και αυτοί οι οποίοι κατοικούν μόνιμα κάπου και οι οποίοι κατόρθωσαν να ενταχθούν και να εγκατασταθούν και αυτό είναι τη αρμοδιότητα των κρατών. Αντιθέτω, οι γινομάδε δεν πιστεύετε πω ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα καθεστώ το οποίο θα είναι ειδικό και το οποίο θα είναι Ευρωπαίοι οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουν μια ταυτότητα. Μα ακούτε, ακουγόμαστε, ακουγόμαστε Μάλιστα, λαμπρά. Νομίζω ότι, γιατί πάλι ότι μιλάμε τζάμπα. Ευχαριστώ. Ε, κατά πόσο πραγματικά αυτοί θα είναι νομάδε ή θα είναι νομάδε οι οποίοι θα κινούνται από χώρα σε χώρα. Τι έχετε να πείτε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. haben viel zu tun. So, Minister. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, προσπαθήστε να τετραγωνίσετε τον κύκλο στις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και πόσο χρόνο έχω πρόεδρε να μου πείτε μέχρι που μπορώ να φτάσω να προσέξουμε από πλευράς χρόνου για την παρέμβαση. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, 11 ερωτήσεις ε, σε αυτό το μείζον φάσμα. Είναι πολλές ερωτήσεις, ο χρόνος πιέζει. 45 δευτερόλεπτα για να απαντήσω σε κάθε παρέμβαση το πολύ πολύ. Θα ήθελα να σας πω στην ενημέρωσή μου αυτή ότι η δομή από πλευρά της Ουγγρικής κυβέρνησης είναι κάπως διαφορετική από εκείνη της ε, συνήθους ε, κυβερνητικής δομής ε, που υφίσταται στην Ευρώπη. Και κάποια θέματα δεν αφορούν ακριβώς το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Άλλοι υπουργοί θα έπρεπε λοιπόν να τοποθετηθούν, για παράδειγμα επαγγελματική κατάρτιση, έρευνα, ε, στρατηγική πολιτική για τους ε, τσιγκάνους. Ε, εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι για παράδειγμα η επαγγελματική κατάρτιση δεν ανήκει στο συγκεκριμένο δικό μου χαρτοφυλάκιο για το οποίο είμαι αρμόδια. Λοιπόν, από πλευρά δομή στην Ουγγρική κυβέρνηση. Τώρα, για τι ερωτήσει σα, μία προ μία θα ήθελα να τι εξετάσω. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, αρκετέ παρεμβάσει αφορούσαν το θέμα αυτό. Θα έπρεπε να συνεχίσουμε τη διαδικασία της διαργασίας της Κοπενχάγης. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το ότι θα έπρεπε νωρίσα ηλικιακά να ξεκινά αυτή η κατάρτιση και επίσης η εκμάθηση γλωσσών. Στόχος είναι να εκτεθούν οι νέοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις ε, όπου θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν και να αποκτήσουν γνώσεις να έχουν έτσι τα προσόντα, τις δεξιότητες ε, ώστε να αναπτυχθούν ε, τα ταλαντά τους, ώστε να είναι εξειδικευμένοι ε, προσοντούχοι εργαζόμενοι στη συνέχεια που θα μπορούν με πολύ θετικό τρόπο να εργαστούν και οπουδήποτε θα ήταν επιτυχής. Αυτό το ίδιο ισχύει και για τις γλώσσες, πράγμα το οποίο αφορούσε μια παρέμβασή σας για την εκμάθηση γλωσσών. Αν θέλουμε να ασχοληθούμε με τη στρατηγική ακριβώς για αυτό το θέμα, αυτό πρέπει να δούμε. Μέσω των πιο ε, σκόπιμων διάβλων και δυνατοτήτων θα πρέπει να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστεί και να ε, τονιστεί η ευρωπαϊκή συνιστόσα στην εκμάθηση γλωσσών ώστε να υπάρξει μια στρατηγική για τις γλώσσες που θα εφαρμόζεται και για την επαγγελματική κατάρτιση και για την γενική εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να μπορούν να μαθαίνουν γλώσσες οι νέοι μας. Το 2009 ήταν το έτος της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Και ως προς αυτό η Ουγγαρία διαδραμάτισε τον ρόλο της όπως της αναλογούσε στο επίπεδο πρέσβεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ίδιος ο Έρνε Ρούμπιχερ ο ε, εφευρέτης, ε, αυτός που επινόησε τον κύβο του Ρούμπικ ε, είχε συμμετάσχει. Η Ουγγαρία ήταν πάντα γνωστή για το δημιουργικό δυναμικό που είχε και εκμεταλλευόταν και το να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση είναι προτεραιότητα για μας. Η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καινοτομία, οπωσδήποτε. 3% του ΑΕΠ θα πρέπει να δαπανώνται από τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μας, μία από τις προτεραιότητες μας. Χρησιμοποιούμε, δρατώμεθα κάθε ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουν τα κράτη-μέλη και να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά τη σπουδαιότητα της επίτευξης αυτού του στόχου. Καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα για την συνδρομή, υποτροφίες και υποστήριξη, διότι όλα αυτά συνδέονται στην έρευνα, στην δημιουργικότητα με την συνδρομή και την υποστήριξη που θα δίνουμε στα πρικισμένα άτομα. Αρκετές κάποιες ερωτήσεις έγιναν όσον αφορά τη στρατηγική για τους Ρωμά, για τους Τσιγκάνους. Στη νέα Ουγγρική κυβέρνηση υπάρχει ένας ολόκληρος θεσμός που μπορώ να πω δεσμεύεται, έχει δεσμευτεί ακριβώς υπέρ της ε, κοινωνικής ένταξης των συγκάνων. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και όχι πρόβλημα ε, εθνοτικής ή εθνικής προέλευσης και ο αρμόδιος ο οποίος θα έχει ε, συνάντηση το απόγευμα θα είναι σε θέση να απαντήσει για την στρατηγική της Ουγγρικής κυβέρνησης ε, και το αντίστοιχο που ακολουθούμε εμείς ε, ως προς την Ευρώπη παρότι υπάρχουν εδώ προβλήματα ε, όσον αφορά την εγκατάλειψη των ε, μαθητών, την ε, αποχώρηση μαθητών πρόωρα από τα σχολεία προτού ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, πρέπει να βρούμε μέτρα και μέσα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτής της ομάδας που μπορεί να θεωρηθεί ως μειονεκτική ομάδα και έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την πολύ έγκαιρη εκπαίδευση των παιδιών, στη σχολική εκπαίδευση, ώστε το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός να μπορεί να έχει πρόσβαση και σε νηπιαγωγεία και σε βρεφ, βρεφονηπιακούς σταθμούς διότι γύρω στην ηλικία των τριών ετών βλέπουμε ότι αναπτύσσονται, έχουν ήδη αναπτυχθεί οι δεξιότητες και οι ικανότητες του λόγου, της ε, απορρόφησης γνώσεων και της μάθησης νέων δεξιοτήτων. Εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν ε, συμμετέχουν σε, σε τέτοιου είδους ε, θεσμούς όπως ε, βρεφονιπιακούς σταθμούς, ε, νηπιαγωγεία, η μειονεξία τους θα αυξηθεί, θα ε, γίνεται όλο και οξύτερη και γι' αυτό πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες όπως δεσμευόμαστε ώστε με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη να τις υιοθετήσουμε και εμείς στην Ουγγαρία και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την πρώιμη παιδεία και εκπαίδευση για τα παιδιά αυτά των συγκάνων. Και το θέμα των ομάδων τσιγκάνων είναι κάπως διαφορετικό ως ε, θέμα. Όμως η στρατηγική για τους τσιγκάνους συνολικά θα πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε αυτό ως ε, ε, παράμετρο. Και όσον αφορά την συνεισφορά μας πρέπει να λάβουμε υπόψη στις δράσεις μας και αυτό. Τώρα, σε σχέση όχι μόνο με την Ουγγρική Προεδρία, αλλά θα έλεγα σε ένα εγχώριο θέμα που έχει ε, επιπτώσει στην Ουγγρική εσωτερική πολιτική, δεν θα ήθελα καθόλου να αποφύγω αυτή την ερώτηση. Να απαντήσω στην κυρία Τρούπελ ότι δεν είχα ενημερωθεί για το γεγονό αυτό εχθέ, διότι βρισκόμουν καθοδόν προ τι Βρυξέλλε. Πρέπει όμω να τονίσω ότι δεν υπάρχει τέτοια αρνητική διακριτική μεταχείριση των συγκανόπουλων, των παιδιών των συγκάνων στην Ουγγαρία. Εκατοντάδε παιδιά πάνε στο σχολείο κανονικά όπως ε, τα άλλα παιδιά ε, που, ε, και δεν έχω ακούσει, δεν έχω πληροφορηθεί για τέτοιου είδους κοινωνικό αποκλεισμό. Αν σημαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες διακριβώσεις και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν θα πρέπει να υποστούν και τις επιπτώσεις της κυρώσεις του νόμου. Δεν έχω όμως ενημερωθεί για αυτό το θέμα, δεν έχω λεπτομέρειες και λεπτομερή γνώση. Όσον αφορά τη σχολή της φιλοσοφίας και την δαπάνη, την ε, ε, χρήση ε, κονδυλίων και όσον αφορά τέτοιου είδους βραβεία. Το θέμα αναφέρεται, έχει αναφερθεί σε δικαστήριο. Δεν αφορά μόνο αυτούς τους φιλοσόφους αλλά και ένα ευρύτερο κύκλο ατόμων που εμπλέκονται σε μια δικαστική τέτοια επίθεση. Δεν είναι λοιπόν επίθεση εις βάρος των φιλοσόφων στην Ουγγαρία αλλά αφορά την χρήση κονδυλίων από τον δημόσιο Κορβανά σε σχέση με τους στόχους ε, που έπρεπε να διέπουν την ε, ε, χρήση τέτοιων κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν σε σχέση με την ενημέρωση που υπήρξε να πούμε ότι δεν είναι αληθής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για επίθεση κατά κάποιων φιλοσόφων ή κάποιας ομάδας ατόμων. Είναι για την χρήση κονδυλίων και βραβείων που δόθηκαν σε κάποιους ε, ερευνητές και που δεν ευθυγραμμίζονται και δεν συνάδουν με τις αρχές που πρέπει να διέπουν ε, τέτοιου είδους βραβεία και έπαθλα. Τώρα, για το θέμα των παιδιών που εγκαταλείπουν τα σχολεία ε, πρώιμα χωρίς να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, τον κύκλο εκπαίδευσης, υπάρχουν διάφοροι λόγοι και αίτια για αυτό το φαινόμενο. Από ό,τι πιστεύω εγώ θα πρέπει να βρούμε τα αίτια, τα πραγματικά αίτια και να επανορθώσουμε την κατάσταση βρίσκοντας τη σωστή θεραπεία. Έχουμε ε, και παιδιά που εγκαταλείπουν το δημοτικό σχολείο και για διαφορετικούς λίγους λόγους. Διαφορετικοί λόγοι βέβαια ε, είναι εκείνοι που κάνουν τα παιδιά να εγκαταλείψουν την επαγγελματική τους κατάτηση, τον κύκλο επαγγελματική τους, επαγγελματικής τους κατάτησης. Έχουμε άτομα που αποχωρούν και από ε, την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους. Πρέπει να βρούμε τους λόγους και τα αίτια γιατί αυτά τα άτομα ε, φεύγουν, φεύγουν από τα σχολεία και πρέπει να βρούμε τις σωστές, ε, τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσει η υλοποίηση των στόχων μας και να μειωθεί το ποσοστό των ε, όσων εγκαταλείπουν τα σχολεία σε κάτω από 10%. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι και το 10% είναι υψηλότατο ποσοστό και αν δείτε και αν, αν εξετάσετε τα αποτελέσματα σε σχέση με τα κράτη-μέλη θα δείτε διαφορετικά ποσοστά. Κάποιες χώρε είναι κάτω από το 10%, Άλλε είναι πάνω από 10%. Η, ίσως η καλύτερη ε, δυνατότητα θα ήταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ουγγρικής Προεδρίας να μπορούμε να συζητήσουμε τότε στο μέλλον ποσοστά 2 ή 3% ως ανεκτά ποσοστά για όσου εγκαταλείπουν πρόωρα τα σχολεία, τον κύκλο εκπαίδευσή του. Για τη συζήτηση όσον αφορά τι βέλτιστες πρακτικέ, σίγουρα πιστεύω θα ήταν το πιο χρήσιμο χρήσιμο, το καλύτερο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ευρωβουλευτή Τόκες που είπε ότι το καλύτερο μέσο για την κοινωνική ένταξη είναι η παιδεία. Και θα ήθελα να τονίσω ότι και να προσθέσω ότι έχουμε σύνθετα ε, ολοκληρωμένα προγράμματα και εγχειρήματα όσον αφορά τις δράσεις μας που ξεπερνούν τα στενά όρια της ε, παιδείας και εκπαίδευσης. Ε, τα προγράμματα για την, ενό... για νεότητα, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, κινητικότητας, όλα συναυτώνται και αλληλοσυνδέονται με αυτό ώστε να καταπολεμηθεί η μειονεξία κοινωνικών ομάδων όπως των συγκάνων. Αν κάποιο παιδί δεν πάει στο σχολείο ή πάει με σχολείο αλλά δεν έχει μια παράδοση οικογενειακή που να συνοδεύει ε, την ε, δραστηριότητα την επαγγελματική και να υποστηρίζει την επαγγελματική ένταξη και δραστηριότητα και δεν έχει αυτό αποτελέσει καθημερινή πρακτική για αυτά τα παιδιά από πλευρά τη οικογένεια, τότε η επίπτωση του σχολείου είναι αποδυναμωμένη. Δεν καταφέρνει πολλά πράγματα. Μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν μπορούμε να δώσουμε κάποια δουλειά στου γονεί, αν μπορούμε να παράσχουμε επαγγελματική κατάρτιση, στέγαση, δυνατότητα να ασχοληθούν και να απασχοληθούν σε ένα επάγγελμα, σε μια θέση απασχόληση οι γονεί. Πρέπει να ανταλλάξουμε βέλτιστε πρακτικέ για να μάθουμε ένα από τον άλλο. Υπάρχουν χώρε που έχουν μεγαλύτερη επιτυχία, έχουν σημειώσει όσον αφορά αυτή την προσπάθεια από ό,τι άλλε. Μπορούμε να μάθουμε λοιπόν ο ένα από τον άλλο, από του καλύτερου. Στην κυρία Παλιαδέλη, θα ήθελα να πω σε σχέση με την ε, εκπαίδευση και τα θέματα τα ανθρωπιστικά Έχω λοιπόν εγώ σπουδάσει όσον αφορά ε, ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες του ανθρώπου. Γνωρίζω λοιπόν το θέμα και ξέρουμε ότι επιστημονικά και η τεχνολογία και τα τεχνολογικά θέματα θα πρέπει να ενισχυθούν. Αν δεν υπάρχει όμως γνώση της ιστορίας και μόνο τεχνολογικά θέματα προωθούνται, αν δεν υπάρχουν τα πολιτισμικά θέματα και ο πολιτισμός στο επίκεντρο, τότε η Ευρώπη θα είναι φτωχότερη. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε λοιπόν τις ανθρωπιστικές σπουδές με κανένα τρόπο στην ανώτατη, στην ανώτατη εκπαίδευση. Θα ήθελα να ζητήσω όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο να αποφύγουμε τις παγίδες. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς στην Ουγγαρία ζητάμε να υπάρχουν μόνο πτυχία όσον αφορά τις, ε, ε, τον επιστημονικό τομέα ε, στις, στην τεχνολογία για παράδειγμα αλλά να έχουμε και την, τα θέματα πολιτισμού και τις ανθρωπιστικές σπουδές, επιστήμες του ανθρώπου που θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Και ένα ερώτημα για την ενεργό στάση των πολιτών την ε, δυνατότητα οι ενεργοί πολίτες να ληφθούν υπόψη. Τι σχεδιάζει λέει η Ουγγαρία. Έχουμε λοιπόν σχετικά προγράμματα στην Ουγγαρία που ε, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά τους στην διάσκεψη που θα διεξαχθεί. Θα είναι μια άτυπη ε, συνάντηση των Υπουργών και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αναφερθούμε και στα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλειών. Πολλοί ε, πραγματογνώμονες, επαΐοντες, καθηγητές θα προσκα... προσκληθούν σε αυτή την άτυπη συνεδρίαση, σε αυτή την διάσκεψη που θα δώσει την προοπτική που θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να συζητηθεί περαιτέρω. Θα είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσουν προγράμματα που θα δρομολογηθούν, που θα είναι γόνιμα, θα είναι καρποφόρα και επιτυχή στην διάχυση πληροφοριών και στοιχείων για την ε, νεότητα και τους νέους να ενημερώνονται περισσότερο για την ιστορία, τον πολιτισμό, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νέοι και να συνεισφέρουν αυτοί οι νέοι έτσι στην ενδυνάμωση της Ευρώπης. Ο ουσιώδης στόχος είναι φυσικά να έχουμε μια ισχυρή, ολοκληρωμένη Ευρώπη που θα ολοκληρώνεται με αυτά τα εγχειρήματα από τους νέους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ την ερώτηση του κυρίου Καβαντά να διαβιβάσετε στον αρμόδιο συνάδελφό σα για να απαντηθεί. Ρώτησε ο κύριο Καβαντά αν προβλέπετε μια πρωτοβουλία για τους νομάδες και αν θα μπορούσε κάτι να γίνει καλό θα ήταν λοιπόν να διαβιβαστεί η ερώτηση να απαντηθεί από τον συνάδελφό σας αρμόδιο. Ελπίζουμε να ακούσουμε κάτι από πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας ως απάντηση αυτή της ε, ερώτησης. Ελπίζουμε για το θέμα των συγκάνων, μια και αυτό ήταν πάντα ένα φλέγον και εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φλέγον θέμα και όσον αφορά την ε, δική σας συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε με την αποστολή της κυρίας Γιαρόκα που είναι εκπρόσωπος των Συγκάνων, ανήκει στην εθνοτική ομάδα των Συγκάνων και ήρθε στην Ευρωβουλή και πρέπει να συζητώνται αυτά τα θέματα όπως αρμόζουν, όπως θα έπρεπε. Και έτσι λοιπόν σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και αυτή την ε, παρουσίαση όσον αφορά και την κυρία Γιαρόκα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ξέρουμε ότι είναι σε καλά χέρια αυτή η υπόθεση με το χαρτοφυλάκιο το οποίο ε, είναι ε, στην δική σας αρμοδιότητα όμως καλό θα ήταν όπως και η κυρία Τρούπελ να ρωτήσουμε σε σχέση με αυτό το γεγονός αυτό το συμβάν αληθεύει ή όχι δεν αληθεύουν όλα τα δημοσιεύματα του DPA για παράδειγμα αλλά αν κάτι συμβαίνει συμβαίνει θα ήμουν πραγματικά ευγνώμων αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε. Και πάλι σε σχέση με αυτό το οποίο είπαμε στον συνάδελφό σας για τα θέματα αθλητισμού, το επαναλαμβάνω, δώστε αγώνα, αγωνιστείτε, ώστε αυτά τα προγράμματα να αποκτήσουν κονδύλια όπως συνάδει, ώστε η στρατηγική 2020 να υποβοηθηθεί και να μπορέσει να ευδοκιμήσει. Δεν θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και δεν θα διέρθουμε από αυτή την κρίση αν δεν έχουμε την καλύτερη παιδεία και κατάρτιση. Περισσότερα πρέπει να γίνουν στο επίπεδο αυτό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σα ευχαριστώ θερμά. Και ίσω καταφέρει, ελπίζω, η Ουγγρική Προεδρία να ε, δημιουργήσει κάποιο ενδιαφέρον και για την Ουγγρική γλώσσα που είναι πάρα πολύ δύσκολη να ε, ενδιαφερθούν περισσότεροι για αυτήν. Ή αναφέρθηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των γλωσσών. Και όταν αναφέρεται αυτό θέλουμε να, είμαστε, να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα ε, για την αναγνώριση αυτή. Θα θέλαμε να ξέρουμε όμω ποιο ξέρει και ποιο μιλάει Ουγγρικά εκτό των Ούγγρων, εκτό Ουγγαρία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε κάτι να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ. Ήταν καλό το ότι επεξηγήσατε ποιοι είναι οι στόχοι σας. Βρισκόμαστε ευθυγραμμισμένοι ακριβώς στην ίδια πορεία. Ευχαριστώ. Επόμενος τώρα θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρος, έχουμε ένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βρίσκει θέση να καθίσει. Λοιπόν, να λυθεί το πρόβλημα παρακαλώ. I see. Inese helps them. Yes. Okay, thank you. Merci, au revoir. Please let them sit where when nobody is sitting. Ο κ. Μπρέντερστροφ, παρακαλώ, καθίστε εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν κενές θέσεις. Στη δεύτερη σειρά. Γιατί δεν, με, δεν έχουν προσέλθει βουλευτές. Εδώ, εδώ η δεύτερη σειρά στους αναπληρωτές. Υπάρχουν πολλές θέσεις για την Κομισιόν κανονικά. Λοιπόν, περνάμε τώρα Συνεχίζουμε την ακρόασή μας. Έχουμε ανάμεσά μας σήμερα τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Σέτς. Ελπίζω να μην το πρόφερα τελείως στραβά το όνομά σας. Όχι. Α, όχι όμως, σωστό. Εντάξει, μάλιστα. Και θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε, πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική, το μελλοντικό έργο των επόμενων έξι μηνών για την Ουγγρική Προεδρία. Ξέρετε ότι έχουμε την έκθεση Σάντσες Σμιτ για το θέμα του πολιτισμού και της ε, συναφούς ε, βιομηχανίας και το θέμα του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις των πολιτισμικών θεμάτων. Έχουμε και την ελπίδα φυσικά επίσης ότι η Ουγγρική Προεδρία τον Μάιο επιτέλους την έκθεση του, της ετικέτα, πολιτισμικής ετικέτας Label λέει η Πρόεδρος θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και δεν θα υπάρξουν δυσκολίες από το Συμβούλιο και έτσι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το Μάιο στην Ευρωβουλή. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο επ' αυτόν που θέλετε να μας εκθέσετε. Tisztelt elnök asszony, Πρόεδρε, και κύριοι, καθώς γιορτάζουμε τα 100 χρόνια μετά το, τη γέννηση του Franz Liszt, πολύ συχνά ακούμε το συμφωνικό ποίημα του που τηλεφορείται Le Prelude. Αλλά πολύ σπάνια ακούμε αναφορές στις ε, ποιητικές περισυλλογές του Αλφόνς Λαμαρτίνς, τον κύκλο των πρελουδίων που ήταν αφιερωμένο στο Βίκτορα Ουγκό και που ενέπνευσε τον συνθέτη Λίστ. Εάν διαβάσουμε αυτό το ποίημα θα δούμε πόσο συμβολικό είναι σε ό,τι αφορά την ιστορία της Ευρώπης και δυστυχώς όχι μόνο στις εποχές του Λαματίν και του Λίστ και ακόμη και μετά στους επόμενους, ε, στα επόμενα χρόνια. Ακούμε τον θόρυβο των 100 στρατιωτών που πορεύονται ως ένα σώμα. Απαγγέλει ο ομιλητής κλπ και η ιστορία της Ευρώπης όπως απεικονίζεται από τον ποιητή και τον συνθέτη με τόσο ευφυή τρόπο και αναφέρεται το 1822 ε, ο ποιητής αλλά δεν ε, ενθυμόμαστε όλοι τις μάχες του επόμενου αιώνα. Για αιώνες λοιπόν η ιστορία της Ευρώπης ήταν μια ιστορία μίσους, ε, στρατών ε, που αντιμάχονται, κυρίως μια ιστορία θανάτων. Θα πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτό κατά τον 21ο αιώνα και το καλύτερο εργαλείο μας είναι ο πολιτισμός. Ίσως να είναι κάπως περίεργος τρόπος ε, να προσεγγίσουμε το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας στον τομέα του πολιτισμού. Αλλά χωρίς μια ιστορική προοπτική δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τους στόχους που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας είναι να σφυριλατήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και να μετατρέψουμε αυτή την Ήπειρο σε Ήπειρο ειρήνης, όπως ήλπιζε ο ε, Εμμανουήλ Καντ στα συγγράμματά του. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό το επόμενο εξάμεινο. Επιθυμούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρία κύρια θέματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Πρόθεση του Ευρωπαϊκού Σήματος για την ε, Πολιτιστική Κληρονομιά, η συνεισφορά του πολιτισμού στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 και κατά τρίτο λόγο προώθηση και ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πολιτισμού και στον οπτικοακουστικό τομέα επίσης έχουμε δύο σημαντικές προτεραιότητες την προστασία των ανηλίκων στις νέες τεχνολογίες και την διαχείριση του ε, δημιουργικού ε, περιεχομένου online. Επίσης θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, ψηφιακή βιβλιοθήκη Ευρωπιάνα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου του Ουγγρικής Προεδρίας. Προγραμματίζουμε να οργανώσουμε 7 συνέδρια εμπειρογνωμόνων και μία άτυπη ε, συνεδρίαση υπουργών. Και επίσης το επίσημο συνέδριο των ε, Υπουργών Πολιτισμού και Παιδείας στις 19 ε, και 20 Μάιου. Θέλουμε να αναγνωριστεί ευρέως ότι ο πολιτισμός διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και ε, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός ότι η ε, πολιτισμική διαφορετικότητα βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτή είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Η αναζωγόνηση και η αναγέννηση και η αλλαγή στην κλασικιστική Ευρώπη ενισχύεται και, και εμπλουτίζεται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς. Η διαφορετικότητα δίνει ένα καλό πλαίσιο στις προτεραιότητες πολιτικής μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν, μου επιτρέψετε, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα τώρα να στραφώ στις προτεραιότητες εν λεπτομέρεια. Τίποτα δεν θα μπορούσε να ήταν πιο συμβολικό από το Ευρωπαϊκό Σήμα για την ε, Πολιτιστική Κληρονομιά. Είναι μια προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία. Η Ουγγαρία ήταν ένα από τα κράτη-μέλη που ξεκίνησαν την διακυβερνητική πρωτοβουλία που αποτελεί τώρα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ε, μια ε, εις βάθος γνώση του πολιτισμού της Ευρώπης μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις ηρωικές στιγμές, τις επιτυχίες, τις αξίες ή ε, τα ανεπίτευτα όνειρα που μας οδήγησαν στο στάδιο που είμαστε τώρα στην Ευρώπη. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να αναλογιστούν τις αξίες που αποτελούν τη βάση της Ευρώπης. Θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να γνωρίσουν περισσότερα για αυτές τις αξίες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους οι νέοι σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και την εθνική ιστορία και κουλτούρα. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για την ενίσχυση της ε, συνειδητής πολιτότητας στην Ευρώπη. Ε, καλωσορίζουμε τα αποτελέσματα της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και ε, πολλά από τα θέματα που γέρθηκαν από το Κοινοβούλιο σας είναι παρόμοια με αυτά που συζητήθηκαν και στο Συμβούλιο. Ω εκ τούτου έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι και να ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα καταλήξουν σε συμφωνία στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Γι' αυτό επιθυμούμε να ε, καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο, αλλά θέλουμε να ε, κάνουμε και πρόοδο στον τομέα της δικτύωσης ή της συνεργασίας ανάμεσα ε, σε ε, σημεία τα οποία είναι υποψήφια. Γι' αυτό ε, στις αρχές Ιουνίου θα έχουμε ένα φόρουμ στο Βίσεγκράτ, στην πόλη του Βίσεγκράτ, για το θέμα του Ευρωπαϊκού Σήματος, για την υλοποίηση των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Σήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και ελπίζουμε το Βασιλικό Παλάτι Ανάκτορο του Βίσεγκρατ που είναι ε, επίση ε, κατέχει το σήμα αυτό θα είναι ένας χώρος που θα εμπνεύσει το φόρουμ στις εργασίες του. Μια άλλη προτεραιότητα πολιτικής κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο ε, κουλτούρα μπορεί να ε, υλοποιήσει τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Η στρατηγική δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στον πολιτισμό ως τομέας που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να κτίσει μια η φορο και ε, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ωστόσο η Ουγγρική Προεδρία είναι πεπισμένη ότι ο πολιτισμός μπορεί όντως να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό Θέλουμε να οικοδομήσουμε πάνω στο έργο που ξεκίνησαν οι προηγούμενες προεδρίες και να εντοπίσουμε τους τομείς όπου ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπης 2020 θέλουμε να εντοπίσουμε εκείνα τα μέτρα, εκείνες τις δράσεις που είναι απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. ο γενικός και φιλόδοξος στόχος είναι να διασφαλίσουμε την σωστή χρηματοδότηση για τον πολιτισμό ε, στο επόμενο ε, ε, πλαίσιο που ξεκινάει το 2014 και ελπίζουμε για την έγκριση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορφής του Συμβουλίου τον, του Μαΐου. Έχουμε τρεις στόχους σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και θέλουμε να δούμε το οικονομικό δυναμικό του πολιτισμού, συγκεκριμένα ε, στους τομείς πολιτισμού και δημιουργικότητας και κατά δεύτερο λόγο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός μπορεί να ενισχύσει το, την κοινωνική συνοχή και κατά τρίτο λόγο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στο να κτίσει μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία. Τώρα, σχετικά με αυτό και σε συνεργασία με την Κομισιόν διοργανώνουμε στις 28 ε, Φεβρουαρίου μέχρι Μαΐου ένα συνέδριο στη Βουδαπέστη και αυτό το θέμα θα τεθεί και στη συνάντηση των υπουργών, στην άτυπη συνάντηση των υπουργών ε, πολιτισμού στις 27 και 28 Μαρτίου. Ελπίζουμε ότι αυτές οι δύο συνεδριάσεις θα μας οδηγήσουν στη τελική διατύπωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Μία προτεραιότητα του Συμβουλίου για το 2011, 12, 13 και 14 είναι προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτισμού. Χάρηκα που άκουσα πόσο σημαντική είναι η κινητικότητα ε, και στα άλλα όργανα και στο Κοινοβούλιο και ο το πρόγραμμα πιλότος που ξεκινήσατε είχε πολύ σημαντικές εμπειρίες. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τα εμπόδια στην κινητικότητα των ε, καλλιτεχνικών εμπειρογνωμόνων και των καλλιτεχνών και θέλουμε να θέσουμε ένα σύστημα ε, πληροφόρησης. Αν ένας καλλιτέχνης θέλει να μετακινηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος για να εργαστεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και από αυτό το σύστημα πληροφόρησης. Και θέλουμε να εγκρίνουμε επίσης τις ε, αποφάσεις, ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου στο επόμενο ε, Συμβουλίο. Το προσχέδιο ενθαρρύνει την κινητικότητα, καθορίζει τους κυριότερους στόχους και τους τρόπους αυτού του συστήματος πληροφόρησης και επιθυμεί να προωθήσει τη διοκτήωση και την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτά θα συζητηθούν στο Συμβούλιο ε, κατά την ε, Ουγγρική Προεδρία για πρώτη φορά και ελπίζουμε να οδηγήσουν σε ένα τελικό έγγραφο. Ο πολιτισμός ε, μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο και στις εξωτερικές σχέσεις μπορεί να αποτελεί καταλήτη στις εξωτερικές μας σχέσεις. Εάν ενσωματωθεί σωστά στις εξωτερικές σχέσεις μπορεί να έχει ε, πολύ θετικό αντίκτυπο συμπεριλαμβανομένου της κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Άρα λοιπόν χαιρόμεθα ιδιαίτερα που βλέπουμε ανάμεσα στις προτεραιότητες την ενίσχυση του ρόλου του, του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις και θέλουμε ο πολιτισμός να ενταχθεί σε αυτό το τομέα των εξωτερικών σχέσεων ε, στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτούς τους πολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση που θα θέσει επιτάπητος ε, ε, θα έχει μάλλον τη συμμετοχή σημαντικών ε, εμπειρογνωμών στο θέμα του πολιτισμού και των πολιτιστικών πρωτεύουσών. Εδώ θέλουμε να συζητήσουμε τον, την πολυπολιτισμικότητα, την πολιτισμική διαφορετικότητα και τις σχέσεις με τις γειτονές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, Κατά ε, την συνάντηση του Συμβουλίου θα γίνει τον Μάιο, θα ληφθεί απόφαση για την πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης του 2015. Αυτά για το θέμα του πολιτισμού. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στην πολιτική των οπτικοακουστικών μέσων. Προτού περάσω όμως αυτό το θέμα, θα ήθελα να υποδείξω ότι η πολιτική αυτή είναι κοινή αρμοδιότητα δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Εθνικών Πόρων, στο οποίο βρίσκομαι εγώ ως και στο δεύτερο Υπουργείο, το Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, που είναι υπεύθυνη για την, τον κινηματογράφο, το πολιτιστικό περιεχόμενο και την ψηφιοποίηση. Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο Υπουργεία ε, είναι πολύ στενή σχετικά με την ψηφιοποίηση και το, την βιβλιοθήκη Ευρωπαίανα, την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ευρωπαίανα είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για, για μας και καλωσορίζουμε τις συστάσεις της ομάδας σοφών που ε, ε, εδώ η νέα αναγέννηση, το, έχω, το διαβάζω από τότε που δημοσιεύτηκε και είναι σχετικά με την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου θα μελετήσουμε αυτές τις συστάσεις και ε, όταν διαβουλευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, δούμε πώς θα προχωρήσουμε με αυτές τις συστάσεις. Ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ισχυρή προστασία των ανηλίκων, ανεξαρτήτως του τύπου μέσων στο οποίο αναφερόμαστε. Τα παιδιά και οι νέοι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες φυσικά αλλά είναι ε, οι πιο τροτές ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα ενεργός στην προστασία των ανηλίκων. Δύο συστάσεις του Συμβουλίου του 1998 και του 2006 μαζί με το Κοινοβουλίο και υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο τομέα αυτό. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι λόγω της ε, ταχείας ε, πρόοδου στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε, να αναθεωρήσουμε τους κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ. Γι' αυτό προσβλέπουμε στις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων του Συμβουλίου του 1998 και του 2006 μετά από την έκθεση της Κομισιόν θα ελπίζουμε να εγκρίνουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου όπου το Συμβούλιο θα καλεί τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις υφιστάμενες συστάσεις και πρότυπα λαμβάνομενων υπόψη των τεχνολογικών αλλαγών. Τέλος, η Προεδρία θα εξετάσει επίσης και την αναγκαιότητα αναθεώρησης ε, των συστάσεων του 2006. Η διαχείριση του online δημιουργικού περιεχομένου είναι ένας άλλος τομέας προτεραιότητας όπου έχουμε δει τρομακτικές άλλαγες. Η ψηφιακή επανάσταση έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε και παράγουμε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα και το εμπόδιο στην ανάπτυξη δύο συνοριακών υπηρεσιών είναι η κατακαιρματοποίηση του ε, ψηφιακού, ε, της ψηφιακής αγοράς. Είναι ε, σαφές αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αφαίρεσουμε αυτά τα εμπόδια που χωρίζουν τα κράτη-μέλη για τις εθνικές αγορές. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια ενιαία ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά. Η Ουγγρική Προεδρία προσβλέπει την Πράσινη Βίβλο που θα δημοσιεύσει το 2011 η Κομισιόν και που θα αναλύει ε, τις δυσκολίες σχετικά με τις δημοσιεύσεις online δημιουργικού περιεχομένου. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις που να εγγυώνται και να διασφαλίζουν την επιλογή αλλά και ε, δίκαιο εισόδημα αυτών που δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο. Είναι περίπλοκο αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε τη στενή συνεργασία ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και της ε, ιστορικής αγοράς. Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε σε αυτό το τομέα εξαρτώνται από το πότε θα ε, δημοσιευτεί η πράσινη βίβλος από την Κομισιόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα οργανώσουμε ένα συνέδριο για το μέλλον του ε, κλάδου αυτού από τις 29 και 30 Απριλίου και θα ε, εστιάζεται στην ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικού κλάδου στην Ευρώπη. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαι πεπισμένος ότι μέσα από τον πολιτισμό και με τον πολιτισμό μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση και την οτροπία των Ευρωπαίων που δεν βλέπουν πλέον την ε, Ένωση ως ε, μόνο οικονομική ένωση αλλά και πολιτισμικό, πολιτιστικό χώρο που μας εμπλουτίζει, που μας ενισχύει που μας κάνει πιο ανοιχτούς. Η Ουγγρική Προεδρία μπορεί να συνεισφέρει και μέχρι το τέλος αυτού του εξαμήνου ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πιο ισχυρή ένωση χωρίς αποκλεισμούς και θα μπορούμε να είμαστε μέρος ε, και θα μπορέσουμε να δώσουμε περάσουμε τις κοιτάλες στους Πολωνούς συναδέλφους. Έχουμε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Έξι έχουμε που θέλουν να παρέμβουν με ερωτήσεις ευρωβουλευτές. Αν παραμείνουμε στους έξι, θα τηρήσουμε το χρονικό όριο. Ο κύριος Καβαντά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τους διάφορους άξονες παρουσίασης της εργασίας σας για την Ουγγρική Προεδρία. Εκτιμώ ιδιαίτερος και δεν είμαι βεβαίω ο μόνος ότι αναφερθήκατε εσείς στον αιώνα του πολιτισμού και της βαρβαρότητας που υπήρξε, που υπήρξε ο 20ος αιώνας. Εγώ στρέφω μεγάλη εκτίμηση στην Ουγγρική κουλτούρα και στο λαό και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από την ιστορία σας ότι θα πρέπει να θυμίσετε αυτό το η βαρβαρότητα. Η Ουγγαρία ε, κατεκτήθη από τους Οθωμανούς, τους Αυστριακούς, τους Ναζί, τους Σοβιετικούς και αρκούμε σε αυτά για να μην μιλήσω και για άλλα. Αλλά μιλήσατε για τον Βίκτορα Ουγκό καθώς επίσης και για τις ελευθερίες τις υποσίες τις οποίες υποστήριξε είστε μέλος της, του κυβερνήσεως αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι του χαρτοφυλακίου σας αυτό το θέμα. Χθε η κυρία Νέλη ζήτησε για μία ακόμη φορά στην κυβέρνηση της Βουδαπέστης να ξαναδεί το νόμο για τα μίντια για να συνάδει με τα βασικά δικαιώματα της ΕΕ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πολύ απλό. Κατά πόσο θα αλλάξετε, τροποποιήσετε αυτό το νόμο ούτως ώστε να συνάδει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και κάτι άλλο το οποίο με εξέπληξε ιδιαίτερο είναι ότι σε μια χώρα όπου ο λαός υπήρξε τόσο θαραλέος στην φορολόγηση των, εξ, ε, ξένων ε, επιχειρήσεων και των πολιτών πραγματικά έχει φτάσει σε τέτοιο ποσό. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω το Ατήλα, τον, τον Κοπάτσι, τον, το Σάντορ Μαράι και τους Καρτές. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα μεγάλα πνεύματα που ήταν Ούγγροι. Πρέπει να αλλάξει αυτό το νόμο κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπαντία Κουτσέτ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις επεξηγήσεις σας εδώ σε σχέση με τις πολιτικές για τα θέματα πολιτισμού. Κάνουμε λόγο για πολιτικές τις οποίες έχουμε μικρές αρμοδιότητες, όμως αντίθετα έχουμε μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες ευθύνες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κάνατε λόγο για ένα στόχο για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινή ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι ταυτότητες δεν μπορούν να δημιουργηθούν πιστεύω εγώ. Είναι συνέστημα, είναι αίσθημα οι ταυτότητες και μπορούν να γίνουν κάποιες ε, δράσεις ε, για πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν κάτι τέτοιο πολλοί έχουμε συζητήσει για την ανάγκη, αυτή την αναγκαιότητα μια ευρωπαϊκή τέτοια ταυτότητα και πολλέ φορέ ακούγονται φωνέ που λένε χρειαζόμαστε αυτή την κοινή ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την προσέγγιση. Όμω το βλέπω πολύ δύσκολο να είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε όλοι σε μια πολιτική ιστορία, κοινωνική ιστορία, κοινή ιστορία τη Ευρώπη. Διότι υπό πολλέ πτυχέ υπάρχουν διαφορέ και διαφορετικά τα βλέπουμε. Και έχουμε πρόσφατε αλλαγέ ε, ιστορικέ που λείπει η ιστορική προοπτική ακόμα σε αυτές. Τα λέω αυτά γιατί δύσκολο θα ήταν να γίνει λόγος για μια αυτή τέτοια ιστορία κοινωνική, πολιτική. Πιθανότατα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θα είναι κοινό και θα είναι κοινή αυτή η ιστορία. Και αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει να δούμε τις ανταλλαγές ε, και τις ε, ε, συσχετήσεις. Κάνατε λόγο για τον Λίστα, για την μουσική, για τι τις καλές τέχνες. Εδώ υπάρχει κοινό χώρος που ίσως θα βοηθούσε να μπορέσουμε να βρούμε μια προσέγγιση για, αυτό, για αυτή την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σα γι' αυτό. Επίση για τα οπτικοακουστικά γίνεται λόγο για δύο θέματα πολύ σημαντικά. Προστασία των ανήλικων online στο διαδίκτυο και για τα καλλιτεχνικά δημιουργικά θέματα στο online, στο διαδίκτυο. Έχουμε τη συζήτηση, έχουμε το πρόβλημα που γνωρίζουμε. Πώ θα βρούμε ένα σύστημα το οποίο θα διατηρεί την ισορροπία μεταξύ τη ανοιχτή πρόσβαση στον πολιτισμό και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα τα πνευματικά του δημιουργού. Είναι μια συζήτηση που στι ίδιε τι χώρε μα δεν συμφωνούμε πάντα απόλυτα επ' αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει όμω να συζητήσουμε για αυτά και να υποβληθούν προτάσει ε, στο τραπέζι. Θα ήθελα να ξέρω πώ θα μπορούσατε να προωθήσετε να είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση αυτά τα θέματα. Και σε σχέση με την προστασία των ανήλικων στο διαδίκτυο, <clears throat> αυτό το θέμα πρέπει να το τονίσουμε. Είναι ακριβώ ένα από τα θέματα που κάθε χρόνο βρίσκεται στο θέμα της ε, διακυβέρνησης ε, της ε, αντιμετώπισης των θεμάτων στο διαδίκτυο. Είναι μια ευκαιρία για το επόμενο φόρουμ. Ένα θέμα, πώς μπορούμε με τις διαρκείς μεταβολές και αλλαγές στις σύγχρονες τεχνολογίες, πώς μπορούμε και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτή η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο να είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Η Helga Τρούπερ, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτη συγκεκριμένη ερώτηση. Όσον αφορά την πρωτοβουλία Ευρωπαϊάνα. η Ουγγαρία ανήκει σε εκείνε τι χώρε που έχουν το χαμηλότερο βαθμό ψηφιοποίηση. Τώρα, υπό την Ουγγρική Προεδρία, θα μπορέσει να γίνει κάτι πραγματικά περισσότερο. Χωρί να επαναλαμβάνω, θέλω οπωσδήποτε την ερώτηση του κυρίου Καβαντά να την υποστηρίξω και εγώ. Και τρίτον, κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι είσαστε υπέρ της πολιτισμικής λέει πολυμορφίας και ποικιλότητα και ότι με την πολιτισμική αυτή πολιτική την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλετε να την κάνετε έναν πολιτισμικό και πνευματικό χώρο και όχι μόνο να είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση και η Νομισματική Ένωση που, στην οποία θα επικεντρωνόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Ουγγρική πολιτική μάλλον ένα διχασμό πολιτισμικών θεμάτων και πνευματικών θεμάτων ε, οδηγεί στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή που υπογράφει ο Βάσλαβ Χάβελ, ο Κόνραντ που ανησυχούν για το άνοιγμα και την ελευθερία και την ε, ελευθεριότητα του λόγου στην Ουγγαρία. Στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα θέματα τα έχουμε συνειδητοποιήσει και οι πολίτες ανησυχούν και πρέπει να σχολιαστούν όλα αυτά. Δεν επαρκεί να λέει κανείς ότι σας ενδιαφέρει η πολιτισμική ποικιλομορφία. Έχουμε πολλές ενδείξεις για αντισημιτισμό που αυξάνεται όλο και περισσότερο στην Ουγγαρία. Εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμού πρέπει να λάβουμε θέση και να τοποθετηθούμε στεναρά επ' αυτών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μπορώ να προσθέσω τη φωνή μου άρρηκτα στις παρεμβάσεις των προλαλισσάντων. Οι εκθέσεις και οι αναφορές από την Ουγγαρία που ακούμε πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικές και ανησυχητικά γεγονότα. Αυτά που αναφέρατε ως στόχους για την ευρωπαϊκή πολιτική που θα έχετε ως Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου, όλα αυτά που μας είπατε και αυτά που ακούμε από την Ουγγαρία όσον αφορά τα πολιτισμικά, διχάζονται. Το ένα παρεκκλίνει από το άλλο. Έχουμε όλο και περισσότερες αναφορές ότι υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης όσον αφορά τους ε, ε, διανοούμενους και υπάρχουν εκστρατείες κιόλα με προσωπικές επιθέσεις εναντίον τους το Εθνικό Θέατρο, λέει, στην Ουγγαρία, που είχε μια παγκοσμιοποιημένη κατεύθυνση όλο και πιο εθνικιστικό γίνεται εθνοκεντρικό και λέγεται και σε σχέση με τους ε, πνευματικούς ε, ε, ηγέτες ότι το αρχείο Γκέρκ Λούκατς έχει τεράστια προβλήματα διότι έχουν διαγραφεί, έχουν, τα κονδύλια έχουν καταργηθεί και δεν υπάρχει καμία τέτοια δράση. Και όταν μια εφημερίδα όπως η γερμανική Die Welt που δεν είναι καθόλου ε, αριστερή, μάλλον του συντηρητικού στρατοπέδου είναι, όταν ιδιαίτερα ανησυχεί για αυτές τις επιθέσεις που γίνονται στην Ουγγαρία και όλο και περισσότερο αντισημιτικές παρεμβάσεις γίνονται με αυτές τις εκστρατείες, είναι σκόπιμο νομίζω και λογικό κάτι περισσότερο να μας πείτε εσείς. Πώς εσείς δηλαδή αυτά τα οποία εμείς ακούμε από την Ουγγαρία και αυτά που εσείς θέλετε να πράξετε ως στόχο Τη ε, της Ουγγρικής Προεδρίας πώς, που σίγουρα μπορούμε να προσυπογράψουμε κι εμείς πώς αυτή η αντίφαση μπορεί να συγκεραστεί πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την αντίθεση ευχαριστώ ο κύριος Λόταρ Μπίσκι έχει τον λόγο και μετά οι άλλοι συνάδελφοι θα περάσουν στη συνέχεια ίσως σε άλλο γύρο ευχαριστώ κύριος Μπίσκι ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Υπουργέ είναι καλό το ότι εσείς ε, αναφέρατε το μεγάλο Ούγγρο καλλιτέχνη Λίστ εισαγωγικά. Είναι και μεγάλος Ευρωπαίος ταυτόχρονα ο Λίστ. Ένα πρόβλημα θέλω να αναφέρω το οποίο συχνά ε, σκέφτομαι. Έχετε ένα μεγάλο οπτικοακουστικό πρόγραμμα και τώρα τίθεται αυτό το ερώτημα. Και ο Γκέρ Λούκατς είναι ο δάσκαλός μου, θεωρώ εγώ, με τα μεγαλοφυή του σφάλματα αλλά και τις μεγαλοφύης ιδιοφύης ιδέες του. Τι θα κάνουμε τώρα τι θα γίνει με εκείνα τα μέρη του πολιτισμού των χωρών της ε, Ανατολικής Ευρώπης που δεν ταιριάζουν σε ένα μαύρο-άσπρο πλαίσιο. Γιάντσο, για παράδειγμα. Άντζεϊ Βάιντα, σκηνοθέτης από την ε, Πολωνία και άλλους. Και, για παράδειγμα, τον Κουρτ Μέτσιχ, έναν ε, γερμανό σκηνοθέτη που έκανε και ταινίες προπαγάνδας αλλά και άλλες που απαγορεύτηκαν. Και άλλοι και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά σκηνοθετών της Ευρώπης, Ευρωπαίοι σκηνοθέτες που, έχουν, ε, που ήταν δημοφιλείς ε, όσον αφορά τους πολίτες μας και είναι και αυτή συνεισφορά υπέρ της, ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτούς τους ενδιάμεσους, ας το πω έτσι, καλλιτέχνες. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με συγκινεί και με κινεί. Και ελπίζω ότι οι Ούγγροι με αυτά τα μεγέθη τα ενδιάμεσα μεταξύ των μεγάλων και των μικρότερων θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Διότι για ένα μεγάλο πολιτισμό θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και τους πιο αντιφατικούς θα έλεγα, λίγο περισσότερο αντιφατικούς εκπροσώπους της ανατολικοευρωπαϊκής ε, καλλιτεχνικής και πνευματικής ζωής μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτισμικών θεμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις τώρα. Παρακαλώ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνθεση των διαφόρων ερωτήσεων. Ο κύριος Καβαδά είπε και έθεσε ένα ερώτημα καλύτερα και συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή, άρα το συμπέρασμά του θα έλεγα πως ε, θα έλεγα ότι δεν συμφωνώ με αυτές καθότι ε, οι ανησυχίες οι οποίες εξφε... οι της Νέλη Κρούτς Επιτρόπου έχω εγώ λεπτομερείς ε, ε ε, παρατηρήσει που έγινε αυτό είναι το νομικό, τρεις παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν σε αυτό το ένα είναι το νομικό το δεύτερο είναι ο ορισμός τι εννοεί δηλαδή και ποιε είναι οι υποχρεώσεις και το, και το τρίτο είναι θέμα καταγραφής υπάρχουν τρία θέματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε αμφισβήτηση αυτά τα ερώτημα θα πρέπει να, είναι, να διευκρινιστούν πλήρως με βάση έναν ορισμό και θα πρέπει να σωματωθούν, να σωματωθούν μέσα στο νόμο περί των μίδια στην Ουγγαρία. Ωστόσο, διαβάζοντας αυτές τις ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί, πιστεύω ειλικρινά πως εξηγούν τους στόχους που εξυπηρετούν, τις επιθέσεις σε πολιτικούς κύκλους και σε κύκλους των μίντια που αντέδρασαν σε αυτή την εισαγωγή αυτού του νόμου στην Ουγγαρία θα ήθελα να διευκρινίσω πως είναι δεν είναι της αρμοδιότητας μας να κάνω δηλώσει επί του θέματος αυτού και αυτό για διάφορους λόγους αλλά ωστόσο θα πω πως αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα απαντήσω έστω συντόμως. Όσον αφορά το ερώτημα πώς θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συνειδητοποίηση θα λέγαμε σε σχέση μια κοινή συνείδηση ευρωπαϊκή, η οποία πραγματικά σπάζονται οι πάντε και ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, θα λέγαμε. Ιστορικά γεγονότα θα πρέπει να είναι πραγματικά οι φορεις αυτών όλων των πραγμάτων και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα στον 21ο αιώνα τι μορφή μπορεί να λάβει. Κατά τη δική μας ανάγνωση υπάρχουν πολλές παραδόσεις στην ιστορία της Ευρώπης, πολύ καλές όλες και στην πολιτιστική παράδοση βεβαίως και ιδιαίτερα με σκοπό να ταυτίσουμε και να φωτίσουμε τις πιο, τα πιο σημαντικά στοιχεία από όλες αυτές θα πρέπει να τις ερμηνεύσουμε, θα πρέπει να τις δούμε και θα έχουμε ε, έχουμε πολλά καλά εργαλεία, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία βεβαίως, στα οποία μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε. προσωπικά εγώ δεσμεύτηκα σε αυτά τα ευρωπαϊκά project και αν με ρωτήσετε πραγματικά για τη θέση την οποία εκπροσωπώ σε σχέση με το γεγονός ότι η Ουγγαρία και τα ουγγαρικά στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπει ε, δεν έχουν γίνει ψηφιακά αυτά τα στοιχεία αυτό χρειαζόμαστε να κάνουμε και αυτό θα πρέπει να και θα χρειαστεί να αλλάξουμε. Και στους επόμενους 6 μήνες θα έχουμε καλύτερη εξέλιξη σε αυτό το θέμα, δηλαδή το digitalize, το ψηφιοποίηση των στοιχείων. Το Στρούμπελ τώρα, σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Στρούμπελ, τελειώσαμε το πρώτο όσον αφορά τη σειρά των ευρωπαϊκών αξιών, την διαφοροποίηση, το ανώμιο τους, τον πλούτο τους. Πράγμα το οποίο είναι ε, ποια μειονεκτήματα δημιουργούνται και πώς η Ευρώπη δημιουργεί σε μερικές χώρες ε, μειονεκτική θέση. Όπως είπατε, ο Κόρατ, Νόντολόσεν και Κόρα, δύο ε, συγγραφείς, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους σαν αφορά για αυτή τη σκίαση των ευρωπαϊκών ε, αξιών για αυτό τον αντισημιτισμό που αναπτύσσεται στην Ουγγαρία θα πρέπει να επιστήσω την προσημίσω ότι ένας από τους μεγαλύτερους ε, ε του 21ου αιώνα έκανε ένα σχόλιο και έγραψε ένα άρθρο δοκίμιο όσον αυτό ο συμμετισμό στην Ουγγαρία. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Αυτός όμως συμπεραίνει ο συγγραφέας πως οι ιδέες και να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην Ουγγαρία και στις, σε πολλές κεντρώς ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μια παράδοση που υπάρχει μια παράδοση αντισημιτικού λόγου λόγου ομιλίας αυτό έπαιξε ένα δευτερεύοντα ρόλο στον πολιτικό λόγο και τα πολιτικά κόμματα τα οποία οικοδομήθηκαν πάνω σε αυτή τη ρητορική πάντοτε βεβαίως έβαλαν και αυτό μέσα και το κόμμα το ΜΥΠ το οποίο απεκλείστηκε από το κοινοβούλιο πριν από χρόνο ήταν μια καλή επίδειξη του μαθήματος αυτού ότι ο αντισημητικός λόγος έδειξε ότι αυτοί που το πιστεύουν πραγματικά και όχι σε δευτερεύοντα λόγο είναι 5% και λιγότερο από 5%. Βεβαίω υπάρχει ε, μια κρυμμένη, ένας κρυμμένος αντισημιτισμός, μια κρυμμένη ξενοφοβία, αλλά από τότε που είναι στην κυβέρνηση η δική μου, το δικό μας κόμμα, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αυξήθηκε ο αντισημιτισμό. Δεν μπορώ πραγματικά να αποσπαστώ κάτι τέτοιο και πρέπει να το απορρίψω ότι υπάρχει αύξηση του αντισημιτισμού. Υπάρχουν σήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν, θα πρέπει να ενευρηθούν, αλλά δηλώσεις και τέτοιου είδους λόγοι, τέτοιου είδους τάσεις οι οποίες υπάρχουν, ότι αυξάνονται, δεν το πιστεύω, κατά την άποψή μου πάντοτε το θέματα του Εθνικού Θέατρου, θέατρου και ορεινών Αρχείων η κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά τη. αμέσως χτυπήσαμε τον κόδωνα του κινδύνου και είπαμε ότι ο διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου θα αντικατασταθεί και θα υπάρξουν και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Οκτώ μήνες πέρασαν και έχω σήμερα μετά 8 μήνες ότι τίποτα δεν συνέβη από όλα αυτά. Ωστόσο είναι γεγονός ότι η χώρα η χώρα ε, η, ε, κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση 8 χρόνια κατάχρησης στο θέμα της πολιτισμού και βεβαίως τώρα υπάρχουν πολύ λιγότερα χρήματα για τα αρχεία διαλύονται ή δεν ενδιαφέρουν πλέον όσον αφορά το θέατρο που είναι ένας θεσμός πολιτισμικός πρέπει να αντιμετωπίσει το κλείσιμο, το ενδεχόμενο κλείσιμο. Με τους συναδέλφους μου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα κοντήρια του προπολογισμού, έχουμε ένα υπουργό, δεν έχουμε υπουργό οικονομικών στην κυβέρνησή μας, αλλά υπάρχει κάποιος που είναι υπεύθυνος για τον προϋπολογισμό και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση και να γίνει αντιληπτό πως η κατάσταση αυτή και νομίζω πως σε αυτόν τον τρόπο απαντώ συνολικά και συνθετικά σε διάφορες ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν. Η κυβέρνησή μου λοιπόν δεν βλέπει την κουλτούρα σαν κάτι το πολυτελές. Δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια η κουλτούρα. Άρα μια χώρα η οποία είναι ευημερούσα μπορεί να αντιμετωπίσει πραγματικά πολύ ευκολότερα την κουλτούρα. Αλλά μια χώρα η οποία έχει, έχει σημαντικά ε, εκτελέσεις ε, ε, εκτελέσεις έργων και κουλτούρας θα πρέπει να αυξήσει και την οικονομία. Έτσι λοιπόν εμείς θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τα τρία αρνητικά στοιχεία που αναφέρθηκαν για την κουλτούρα και Κάποιο είπε ότι μπορεί να είναι μέσο, μερικοί μάλλον λένε ότι είναι μέσον προπαγάνδα η κουλτούρα. Η κουλτούρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροποποιηθεί η ταυτότητα μία χώρα, ενό έθνου ή να αλλάξει. Ή άλλοι θεωρούν ότι η κουλτούρα είναι η διασκέδαση και ο πολιτισμό. Και το οποίο βεβαίω είναι όπω και το προηγούμενο. Εμεί καταλαβαίνουμε την κουλτούρα σαν κάτι, ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να παράγει. Έτσι λοιπόν οι πολιτικοί καταλαβαίνουν πολύ καλά οι πολιτικοί, όχι μόνο στην Ουγγαρία, σε όλη την Ευρώπη, α, ότι η κουλτούρα είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που προανέφερα, είναι ένα φαινόμενο και ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά και ελπίδα για τη βελτίωσή της βεβαίως όταν υπάρχει χρηματοδότηση σε καλύτερες συγκυρίες στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε κύριος το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι κάνατε μια έκθεση πάρα πολύ τεράστι, με τεράστιο ενδιαφέρον Πολλέ από τι ερωτήσει που ήθελα να διατυπώσω διατυπώθηκαν από του συναδέλφου μου όπω από την Μαρία Μπαδία για την ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα. Είναι σημαντική αυτή η συνιστόσα μέσω των θεμάτων των πολιτισμικών. Κάνατε λόγο για τον ευρωπαϊκό θησαυρό πολιτισμού που έχουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ όχι μόνο στο θησαυρό που πρέπει να προστατέψουμε αλλά και στο σημερινό πολιτισμό και τον μελλοντικό πολιτισμό ω ταυτότητα τη Ευρώπη. Πρέπει να προδεύσουμε και να μην παραμείνουμε μόνο στην προστασία κάποιου παροχημένου ή παλαιότερου ας το πω έτσι, πολιτισμικού θησαυρού. Και αυτό είναι τα νέα μέσα ε, επικοινωνίας, ο πολιτισμός online στο διαδίκτυο, η συνιστόσα του πολιτισμού μέσα από το διαδίκτυο, ε, ο τρόπος να αντιστοιχούμε τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι αναγκαία για την προστασία αυτού του νέου πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών. Υπάρχει ένα θέμα που αναφέρθηκε που είναι σημαντικό, η κινητικότητα. Η κινητικότητα των διαφόρων καλλιτεχνών. Εδώ ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις συγκεκριμένες. Οι καλλιτέχνες πολλές φορές εξορισμού είναι ε, ενδιάμεση και έχουν δυσκολία να έχουν επαρκή προστασία που είναι αναγκαία και στην ίδια κινητικότητα. Ένας μουσικός που πάει από μια ουγγρική ορχήστρα σε μια ισπανική ορχήστρα μέσω της κινητικότητας. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές δυσκολίες επίσης όσον αφορά την κοινωνική προστασία. Έχετε κάποια ιδέα από πλευρά της Ουγγρικής Προεδρίας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Καλό είναι, σύντομες να είναι η ερωτήσει. Η κυρία Σάντσε Σμιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την άλυση του, για τις διάφορες πτυχέ της κουλτούρας στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Θα αναφερθώ σε δημιουργικές εκείνες επιχειρήσεις η οποία από τη δική μας επιτροπή και η οποία μπορεί να συμβάλλουν στους στόχους, τους οικονομικούς και της ανάπτυξης της στρατηγικής ΕΕ για τα 2011-2014. Είναι παράγοντας συνοχής κοινωνικής και προόδου διαφοροποίησης της κουλτούρας και καινοτομίας. Το βασικό μου ερώτημα λοιπόν αφορά την ανάπτυξή τους, πώς μπορεί να, να απελευθερωθεί τη δυνατότητά τους, η δυναμική τους, τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εμπληφθούν, τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά μέσα, ο, με το, ο συνεταιρισμός με τις δημόσιες αρχές, τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η προσέγγιση της Ουγγρικής Προεδρίας για αυτό το τεράστιο θέμα που εκπροσωπεί αυτές τις επιχειρήσεις, τις δημιουργικές και τις πολιτισμικές, πώς ακριβώς θέλετε να γίνουν αυτά τα πράγματα και ποια πρόοδος μπορεί να γίνει στην ΕΕ. Ευχαριστώ. Η κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, Υπουργό για την πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσίαση και το σχολιασμό του για θέματα που υπερβαίνουν τα όρια ίσως πρακτικών ζητημάτων. Ε, δεν θα μιλήσω εδώ για το ε, ε, σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κληρονομιάς, γιατί το αφήνω ως κομμάτι των διαπραγματεύσεων που θα κάνουμε στη συνέχεια. Επομένως δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου εδώ, θα δούμε πώς θα τα καταλήξουμε ε, σε ένα τελικό κείμενο που θα υποστηρίξει τον μέγιστο στόχο του, που είναι η Ευρωπαϊκή Συνοχή ε, η ερώτηση που θα ε, έχω να κάνω μια παρατήρηση. Α είμαστε ειλικρινεί. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση ούτε να ορίσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αρχαίο και σύγχρονο, ούτε πολύ περισσότερο να ορίσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Την αναζητούμε. Χρειάζεται πολλή δουλειά μέχρι ότου την κατακτήσουμε. Ε, επομένως, με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι η συμβολή της Προεδρίας σας ε, προς την ε, κατεύθυνση αυτή ε, η αναζήτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας αν θέλετε και ο ορισμός της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας θα ήταν μεγάλη με δεδομένο όσα είπατε προηγουμένως για όσα συμβαίνουν στην χώρα σας για ζητήματα όπως έχεις με το θέατρο και τους Ρωμά σε μια άλλη περίπτωση κλπ η ερώτηση που έχω να κάνω είναι πώς μπορούμε με όλα αυτά τα δεδομένα και με όλες αυτές τις δυστυχώς τις ε, διαπιστώσεις να χρησιμοποιήσουμε το, πώς σκοπεύετε εσείς να χρησιμοποιήσετε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ως εργαλείο για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Ευχαριστώ. Τάκουλα. Τάκουλα παρακαλώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό γιατί έκανε μια ευρωπαϊκή παρουσίαση, ήταν πλήρης και έφυξε τα περισσότερα ευρωπαϊκά θέματα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να βρεθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία θα είναι κοινή κάτι το οποίο θα είναι στη που θα πάει, στην Κοπενχάγη και αλλού. Είναι κάτι το οποίο δεν θα βρούμε ε, ούτε στη Νέα Νέα Υόρκη, ούτε στη στη Μόσχα. Υπάρχει ένας τέτοιος σταθμός παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μια, ε, μια τέτοια αποφασιστικό κίνημα προς αυτή. Υπάρχει αυτή η παράδοση η ιουδεο-χριστιανική. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει την Προεδρία τη ΕΕ και αν σκεφτούμε πραγματικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια επίπτωση επί της ευρωπαϊκής κοινωνίας στον τομέα το πολιτιστικό, πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τα πράγματα και πώς ακριβώς μπορούμε να πάρουμε τα σωστά βήματα προς τα, προ, ε, προς τα μπρος όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της δημιουργίας, της δημιουργικότητας η οποία θα πρέπει να, να, αναπτυχθεί και ένα θέμα ηθικό που τίθεται, μια ηθική ισορροπία, πώς ακριβώς θα το δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα του αντισημιτισμού για παράδειγμα, το οποίο τέθη στην ΕΕ, είμαστε κατά του αντισημιτισμού Σήμερα το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπάρξει μια μια, ένας εορτασμός, ένα μνημόσυνο αν θέλετε όσον αφορά τα, τα θύματα του ολοκαυτώματος και θα υπάρχουν πολλοί ομιλητές. Είναι περίεργο λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια να λέγεται πως η Ουγγαρία τα πράγματα ε, έχουν αλλάξει και δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε το παν για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου του αντισημιτισμού. Πράγμα το οποίο με, με ενοχλεί σε αυτή την όλη συζήτηση είναι ότι εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτή την κυβέρνηση της Ουγγαρίας ενώ μαζί θα έπρεπε να συνεργαστούμε και να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Είπατε προηγουμένως πως υπάρχουν ερωτήσεις πολλές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και οι οποίε δεν ανταποκρίνονται στι ειδικέ αρμοδιότητε. Ωστόσο, είναι θέματα τα οποία μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ, άσχετα αν είναι στο χαρτοφυλάκι σα ή όχι. Πολιτικέ οι οποίε ε, θέλουν, οι πολιτικοί με όμικρο γιώτα, θέλουν να, κατα... να καταπολεμήσουν την Ουγγρική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως αυτή η υπόθεση μπορεί να μπει κατά μέρο και η Κομισιόν μπορεί να ρυθμίσει αυτό το θέμα με την Ουγγαρία και για μας θα ήταν πολύ καλύτερο να κάνουμε το πάνω ούτε, ώστε τα 27 κράτη να συνεργαστούν. Πρόεδρε, θα ήθελα να υπογραμμίσω όλα αυτά τα οποία μας είπα και κατά την άποψή μου πολύ συχνά εμείς δείχνουμε ως ευρωβουλευτές βάζουμε τις προεδρίες σε δύσκολες καταστάσεις, ενώπιον δύσκολων καταστάσεων γιατί υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους ενώ υπάρχουν πολύ καλές παρουσιάσεις, παρουσιάσεις οι οποίες συνάδουν με την Ευρώπη και αυτές η Ουγγρική Προεδρία έχει μεγάλους στόχους, θα ήθελα να την υποστηριχθούμε να τις υποστηρίξουμε και να ενισχύσουν πολύ περισσότερο την Ευρώπη στο επίπεδο του πολιτισμού και της κουλτούρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφος Μάρτιν. ναι. Κάπως διαφορετική θέση θα ήθελα να υιοθετήσω από τον προλαλήσαντα. Κύριε Υφυπουργέ, για θέματα πολιτισμού θα ήθελα να στραφώ και να μιλήσω στη συνείδησή σας, να σας συγκινήσω. Μην με διακόπτετε πρόεδρε σας παρακαλώ. Ίσως θα έπρεπε να πάτε και εσείς στην Ουγγαρία. Για διάφορους λόγους δεν μπορώ να βρω κάποια εξήγηση. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτή. Ξέρετε, ακριβώς στον τομέα που εσείς εκπροσωπείτε, μία απάντηση νομίζω όσον αφορά και την αντιπροσωπεία της Κίνας που πάμε στο Πεκίνο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρεμβαίνουμε σχετικά. Τι γίνεται λοιπόν. Εδώ οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι και οι πολίτες εδώ για όποιον ανήκει στους διανοούμενους συγκινεί ιδιαίτερα αυτή η παρέμβαση, παρέμβαση σε σχέση με την τοποθέτηση αυτή από πλευρά σας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου και μάλιστα μια ευρωπαϊκή ταυτότητα κιόλα. Εγώ ίδιο ήμουν μέλος στην Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων και ξέρω πόσο τα θέματα επικέντρωση των θεμάτων ιδιοκτησία του τύπου των ΜΜΕ μας συγκινούν. Αλλά η τέταρτη εξουσία να να εξουδετερωθεί μέσω ενός τέτοιου νομοθετήματος όπως αυτού που εσείς στην Ουγγαρία νομοθετήσατε νομοθετήσατε πουθενά δεν φαντάστηκε κάποιος να δράσει με αυτόν τον τρόπο και δεν το έκανε αυτό. Και στον δικό σας τομέα που είναι ένας κλασικός τομέας ε, και σε σχέση με την αυστριακή κυβέρνηση ε, που είχε προσφερθεί ακριβώς η πολιτική διασύνδεση να μην ε, την χάνει μια υπεκφυγή ότι δεν είναι δική σας λέει αρμοδιότητα και δεν μπορείτε εσείς να απαντήσετε. Να δραστηριοποιηθείτε ώστε από πλευράς Ουγγαρίας να δοθεί μια σαφής απάντηση, μια σαφής τοποθέτηση για τη συζήτηση που έγινε την προηγούμενη Ολομέλεια, την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν ο αρχηγός της κυβέρνησής σας, ο κύριος Όρμπαν, αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία επικρίσεων των Ευρωβουλευτών που μέσα από όλε τις κοινοβουλευτικές ομάδες διατυπώθηκαν, κυρία Πρόεδρε, για αυτή την πρακτική στην Ουγγαρία, για αυτή τη στάση της Ουγγρικής κυβέρνησης, απέρριψε τις επικρίσεις λέγοντας ότι δεν μπορεί λέει, να προσβάλλεται ο Ουγγρικός λαό με αυτόν τον τρόπο. Ήθελε να παρουσιαστεί ως προστάτης του Ουγγρικού λαού και όχι να πει ότι ήταν δική του ευθύνη αυτό. Ζητώ από εσά σαφή τοποθέτηση. Είναι ένα θεμητό πλαίσιο συζήτηση όταν υπάρχει επίκριση για συγκεκριμένο νομοθέτημα να, το συνδέετε, να συνδέετε αυτή την επίκριση με την εθνική σα υπερηφάνεια και να λέτε ότι προσβάλλεται ο λαό λαός διότι εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με αυτά τα θέματα όπω και τον Γιώργη Κόνραντ που έχει υπογράψει μια επιστολή που λέει είναι μια νέα μορφή δικτατορία. Έτσι τοποθετούμαστε. Εσείς τι λέτε. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Μαρτίν αναφέρθηκε στην πρόταση με την οποία ήθελα να ξεκινήσω. Φοβάμαι επίσης ότι δεν θα αφήσουμε το εθνικό το έθνος της Ουγγαρίας να τύχει ε, κατάκριση από γενικευμένε δηλώσεις που ακούστηκαν σήμερα, για παράδειγμα κατηγορίες αντισημιτισμού. Αυτή, αυτά είναι πολύ οδυνηρά. Ε, αυτή είναι πολύ οδυνηρή όρη Από φιλελεύθερη άποψη, αν, αν δεν υπάρχουν ε, επιχειρήματα, τότε πάντα ε, τίθεται το θέμα του αντισημιτισμού. Θα ήθελα να απορρίψω αυτό το πράγμα, διότι στην πρώτη διακυβέρνηση Όρμπαν ήταν η πρώτη που ε, διακήρυξε την ημέρα του ολοκαυτώματος ως ε, επέτειο και η κυβέρνηση ε, πήρε αρκετά μέτρα για να απορρίψει αυτή τη δήλωση. Είναι ένα οδυνηρό θέμα, είναι μια οδυνηρή δήλωση που θέλω να την απορρίψω εδώ. Ο κύριος Τέκες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι λίγο περισσότερο υποκειμενικός. Εγώ γεννήθηκα στην ίδια πόλη με τον Υπουργό, το, στο Κλούζ, Κόλσβαρ, ονομάστε το όπως θέλετε και αγωνιστήκαμε κατά ε, της ίδιας ε, δικτατορίας του Τσαουσέσκου στη δεκαετία του 80. Και πάντα μας ε, κατονόμαζαν αντιρουμάνους και είναι μια παράδοση που έχει επιβιώσει μέχρι και σήμερα. Όταν εξελέγει ευρωβουλευτής, κάποια άλλα μέλη αυτού της Ευρωβουλής με αποκάλεσαν αντιρουμάνο. Αλλά θυμάμαι ότι καταφέραμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους Ρουμάνους φίλους στις κοινούς μας αγώνες κατά της δικτατορίας του Τσαουσέσκου. Αυτά τα θυμάμαι όταν ε, ακούω για αντισημιτισμό και υπάρχει μια διαδικασία δικαστική για την κατάχρηση των ε, ε, δημοσίων κονδυλίων και είναι πολύ εύκολο να φωνασκεί κανείς και να λέει τι είναι αντισημιτισμός. Αν είναι ένας Ρωμά που κλέβει δημόσια χρήματα ή ένας Εβραίος ή Ούγγρος ή όλοι πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου για κλοπή. Όχι γιατί είναι Ρουμάνοι, Εβραίοι, Ρωμά, αλλά γιατί έκλεψαν χρήματα. Γι' αυτό είναι δύσκο, ε, επικίνδυνο να φωνάζει κανείς ότι είναι αντισημιτικό. Και δεν... Ε, εδώ δεν πρόκειται περί ακρόασης στην Επιτροπή Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ επιτρέψτε μου τώρα να ζητήσω να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Παρακαλώ. Um, uh, Προσέξτε, θα ήθελα να, με αντίστροφη σειρά να προσπαθήσω να απαντήσω. Παρατηρήσεις του Hans Peter Martin και του φίλου μου κύριου Τεκέσ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις δεν ήθελα να κάνω λόγο για αυτά τα θέματα. Όμως το γεγονός ότι αν υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα που πραγματικά διακύβευσε πολλά και έδωσε μεγάλες μάχες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παράλληλα προς τον κύριο Τέκες, πρέπει να πω ότι εγώ θα ήμουν το δεύτερο άτομο στις μάχες στους αγώνες αυτούς. Κάποιος ε, με ρώτησε γιατί δεν έχω μία γραβάτα, δεν φοράω παπηγιόν γραβάτα και απάντησα στην ερώτηση αυτή με την ιστορία ότι οι πράκτορες της Σεκουριτάτε ήθελαν να με στραγγαλίσουν με την ίδια μου τη γραβάτα. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος και δεν φοράω πια γραβάτες από τότε. Πραγματικά λοιπόν είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος ε, για αυτά τα θέματα η ελευθερία του εκφράζεστε, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία, οι ελευθερίες αυτές του εκφράζεστε και του λόγου βρίσκονται ακριβώς ε, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου και είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος ε, όσον αφορά τις θεμελιώδεις αυτές αρχές και αξίες. Έχω σταδιοδρομία και επιδόσεις ε, σχετικά. Στην Ουγγαρία όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τα παράγωγα δικαιώματα δεν βρίσκονται με κανένα τρόπο ε, εν κινδύνο. Δεν διακυβεύονται με κανένα τρόπο. Δεν μπορώ να χρησμοδοτήσω βλέποντας σε, σε μια κρυστάλλινη, εξετάζοντας την ε, κρυστάλλινη σφαίρα. Έχουμε όμως ένα νομοθέτημα για τον τύπο. Με διαφορετικό τρόπο μπορούν να ερμηνευθούν πολλά πράγματα. Το Σύνταγμα, τον είπα, δεν θα ήταν επαρκής εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για παράδειγμα, σε, χώρες, σε τριτοκοσμικές χώρες. Και βλέπουμε ότι το γράμμα του νόμου αυτού, δεν αποτελεί εχέγγυο, δεν είναι καμιά εγγύηση από πλευράς του. Και τα πράγματα αποδεικνύονται στην ίδια την καθημερινή ζωή και χρήση πως έχουν πώς τα πράγματα εξελίσσονται. Μόλις ε, υπάρχει γνώση για οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση θεμελιωδών ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα είμαι άμεσα στη διάθεσή σας και θα είμαι πρόθυμος να τα εξετάσω αυτά. Δεν μπορώ όμως να στρέψω, να απεμπολίσω το παρελθόν μου και την ε, δική μου ζωή και την δική μου ηθική και τις αξίες μου. Δεν πρόκειται να απεμπολίσω αυτές τις αξίες. Και φυσικά πολλά πρέπει να πράξουμε ακόμη και στην ίδια την Ουγγαρία, εμείς οι ίδιοι. Από την άλλη πλευρά, από πλευρά των νομοθετών της ίδιας της κυβέρνησης, μέχρι τα πιο διαφορετικά διαστρώματα, στρώματα του πληθυσμού. Έχουμε πολλά να κάνουμε, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολλά πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ετικέτας για προϊόντα πολιτισμικά Νομίζω ότι με αυτές τις προσπάθειες και για την ε, υποστήριξη της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των ε, όσων εμπλέκονται στην καλλιτεχνική ζωή είναι μια δέσμη πρωτοβουλειών και εγχειρημάτων που δεν είναι η ε, εγγύηση αυτών απλά και μόνο για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας αλλά είναι στοιχεία αυτής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, πώς μπορούν οι αρχές αυτές να αποκτήσουν σάρκα και οστά, πώς τα ωραία λόγια θα γίνουν πράξη. Το να σφυριλατήσουμε και να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή κοινή ταυτότητα για τα πολιτισμικά είναι ο τελικός μας στόχος. Η πορεία όμως, η οδός που θα οδηγήσει προς την επίτευξη αυτού αυτού του στόχου είναι μακρά και θα είναι δύσκολη πράγματι. Και ακόμη και οι διαφορετικές ευρωπαϊκές ταυτότητες είναι πολύ ανομοιογενείς. Ας παραμείνουμε στο παράδειγμα του Franz Liszt, μουσικού αυτού. Οι περισσότερες συνθέσεις του Liszt αλλά και του Brahms, Brahms επίσης έχουν τις ρίζες τους στη μουσική των συγκάνων η Ουγγρική, ο Ουγγρικός πολιτισμός αφομοίωνε πάντα και ολοκλήρωνε εντάσσοντας τον πολιτισμό αυτό στοιχεία άλλων. Αυτό είναι κάτι θεμελιώδες αν δει κανείς και τη δουλειά που έκανε ο Μπέλα Μπάρτοκ, ένας άλλος σημαντικός μουσικός συνέθεσε ε, <clears throat> μελήματα τα οποία ενέτασαν και ρουμανικές μελωδίες σε αυτό το ουγγρικό πλαίσιο συνθέσεων που δημιούργησε. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστά ως τελικό προϊόν ουγγρικό. Έχουμε λοιπόν μακρά πορεία και δύσκολη, δυσχερή πορεία που θα πρέπει να διανύσουμε, όμως ξεκινήσαμε αυτή την πορεία προς αυτό το στόχο, βήμα προς βήμα θα προχωρήσουμε. Δεν είναι φυσικά μικρά βήματα αυτά για τους καλλιτέχνες και τους πραγματογνώμονες, διότι είναι σημαντικά τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων, αν μπορούν να υπάρχουν, αν μπορούν να διασφαλίσουν την κοινωνική τους ασφάλιση, σημαντικό θέμα για την ασφάλεια της διαβίωσής τους. Είναι μικρά βήματα για την Ευρώπη, όμως σημαντικά βήματα για τους ε, καλλιτέχνες. Αυτή είναι η πορεία την οποία θα πορευτούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Κυρία Τρούπερ, θέλατε μια ερώτηση να διατυπώσετε, αλλά κανονικά έχουμε ολοκληρώσει. Μια προφορική δήλωση θα κάνω, Πρόεδρε. Είναι τεράστια σημασία. Θέλω να στραφώ στον συνάδελφο Μπάγκο. Όταν έκανα λόγο για το ότι υπάρχουν πολλές μελέτες και άρθρα που λένε ότι συνολικά όλο και περισσότερα <clears throat> αντισημιτικά κύματα σημειώνονται στην Ουγγαρία, αυτό το διαπιστώνουμε από διάφορες ε, μελέτες. Όμως αυτό το οποίο δεν έκανα και βάβω, δεν έκανα προσωπική επίθεση σε κανέναν και δεν τον κατηγόρησα ως αντισημίτη και αυτό είναι διαφορά σημαντική. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσετε αυτό. Εγώ δεν θέλω θέλω με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι προσέβαλα κάποιον. Δεν προσέβαλα κανέναν. Ανέφερα μόνο κάποιες τάσεις που υπάρχουν στην Ουγγρική κοινωνία, όπως αναφέρω αυτές τις τάσεις όταν υπάρχουν και σε άλλες κοινωνίες. Θα ήμουν πραγματικά ευγνώμων αν λαμβάνατε υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση. Μπορώ, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ, απαντά στην Πρόεδρο. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την παρέμβαση της κυρίας Τρούπερ της κυρίας Χέργε Τρούπερ και να πω έχω μια ερώτηση προς εμάς κυρία επίσης Γνωρίζετε την ύπαρξη μιας μελέτης η οποία ενδεικτικά αναφέρει, εμπεριέχει την ανάπτυξη για το φαινόμενο της διάχυσης και ανάπτυξης του αντισημιτισμού ως φαινομένο στην Ουγγαρία ή συγκεκριμένα τους τελευταίους 8 μήνες διότι θυμάμαι ότι είχα διαβάσει στις εφημερίδες περίπου πριν από ένα χρόνο σχετικά ότι ο Γιόμπικ θα είναι λέει ο πιο στενός σύμμαχος του κόμματο Φίντες. Αν έχετε εξοικειωθεί με την εσωτερική πολιτική ζωή στην Ουγγαρία, θα ξέρετε ότι ο Γιόμπικ δεν είναι καθόλου σύμμαχος, αλλά είναι αντίπαλο και ένας από τους πιο επίφοβους αντιπάλους ή ανταγωνιστές του κόμματο Φίντες. Φυσικά υπάρχουν αντισημιτικές τάσεις και υπάρχουν ε, φαινόμενα αντισημητικών λόγων που ε, αναδύονται και εκφωνούνται στην Ευρώπη. Όμω δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τη δική μα κυβέρνηση που έχει θητεία 8 μηνών μόλις ε, στην Ουγγρική κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να υφίσταται λέει αντισημιτικό φαινόμενο στην Ουγγαρία. Στην πολιτική μας για τον τύπο και για τα πολιτισμικά θέματα αυτή η κυβέρνησή μας θέλει να ε, θέσει τα θεμέλια για ένα πραγματικό ευρωπαϊκό λόγο που θα εκφέρουμε και που θα υλοποιήσουμε. Αυτό είναι στόχο μα. Από κοινού με εσά, από με όλε τι πολιτισμένε ε, ε, πολιτικέ δυνάμει στην Ουγγαρία, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και ήδη σα έδωσα κάποια λίγα παραδείγματα. Αν υπάρχει κάποια δύναμη που μπορεί τον, την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό, να, τα, τα προαγάγιος φαινόμενα είναι οι δυνάμεις ε, που προανέφερα εγώ. Είναι οι δυνάμεις ε, αυτές ε, που είναι αντίπαλοι μας, μόνο εμείς και οι σύμμαχοί μας μπορούμε να αντιπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όμως να δείξετε υπομονή και αντοχή και το κάνατε αυτό. Εσείς ως Υπουργός Πολιτισμού είσαστε επίσης υπεύθυνο για τα θέματα τα πολιτισμικά, την ελευθερία του τύπου, ακόμα και αν δεν είσαστε ο αρμόδιος ε, πολιτικός, ε, ε, σε πολιτικό επίπεδο υπουργό για αυτά τα θέματα, ανήκουν στο πολιτισμικό, πολιτιστικό πλαίσιο και πρέπει να αντέξετε και να ανεχθείτε να τα αναφέρουμε εμείς. Θα ήθελα να πω, δεν το βρίσκω καλό, όλο και πιο συχνά να μετράμε και να σταθμίζουμε με δύο μέτρα και σταθμά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε νόμους για τον τύπο που κανείς ωστόσο δεν άσκησε επικρίσεις επ' αυτών. Εντάξει, έχουμε νομοθετήματα νόμους για τον τύπο και ως Προεδρία του Συμβουλίου Κανείς δεν ρώτησε τους Σλοβαίνους οτιδήποτε για τον νόμο για τον τύπο που έχουν. Και ρωτώντας θα μπορούσε κανείς να έχει μάθει κάποια πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να μην υπερβάλλουμε και να μην ξεπερνάμε τα εσκαμένα όταν γίνεται λόγος για κάποια πράγματα. Ο Πρωθυπουργό επίσημα ανέφερε ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γνωμοδότησή τη διαπιστώσει ότι είναι ελληματικό αυτό ο νόμο, τότε θα αλλάξει αυτό το νομοθέτημα. Α αναμείνουμε λοιπόν λίγο μέχρι ότου υπάρξει αυτή η γνωμοδότηση των νομομαθών των επαϊόντων τη Νομική Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω μεγάλη κατανόηση, αλλά είμαι κατά των καταδικών και κατά τη καταδικαστική, ε, καταγγελτική, καταδικαστική προσέγγιση και σε άλλους ε, που έχουν ίδια προβλήματα δεν έχουμε υιοθετήσει άλλη στάση. Θα ήθελα να πω όταν είχε ε, τεθεί υποκύρωση και υποδίωξη η ουγγρική γλώσσα στη Σλοβακία πού βρέθηκαν τότε όλοι αυτοί που σήμερα υποτίθεται ότι είναι υπέρ των μειονοτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των περιθωριακών και μειονοτήτων. Πάντα με τα ίδια μέτρα και σταθμά πρέπει να σταθμίζουμε και να κρίνουμε και όχι κομματικά με ιδιοτέλεια και εξυπηρετώντα προωθώντα δικού μα σκοπού. Με τον κύριο Μάρτιν στην ε, κοινή συνεδρίαση, όπου με την Πολιτισμική Επιτροπή και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και με την Έλλη Κρού είχαμε συνέρθει, σημαντικέ ερωτήσει θέσαμε, που για μένα είναι τεράστια σπουδαιότητα και για όλου μα. Πού πάνε τα πράγματα με το, τις, τις δημόσιες ε, ε τηλεοπτικές αρχές ε, της Ουγγαρίας. Υποστηρίζονται ή όχι, θα μπορέσουν να επιβιώσουν ή όχι εκεί στη χώρα σας. Είναι σημαντικότατα ερωτήματα αυτό και γι' αυτό κάναμε την έκθεση έκθεση Μπέλετ. Εμείς, και το λέω αυτό, πριν από δύο χρόνια, από την Ουγγαρία την ίδια μας το επεσήμαναν αυτό το πρόβλημα. Τότε δεν υπήρχε αυτό το νομοθέτημα για τον τύπο. Μας είχαν πει να εξετάσουμε και να ασχοληθούμε με την κατάσταση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνικών σταθμών στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Αυτό ήταν ο λόγο για τον Μπέλετ. Όχι το νομοθέτημα για τον τύπο τώρα. Όταν έχετε αυτό το νόμο για τον τύπο και τα μέσα ενημέρωση και που διαδέχεται την κομμουνιστική νομοθεσία που ίσχυε μέχρι τότε, ε, πρέπει να ασχοληθούμε για αυτό το θέμα και να δούμε τι θα γίνει. Να μην χάσουμε το καλό ρίχνοντάς το και αυτό με τα αρνητικά στο ΚΕΑΔΑ. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε πραγματικά εμπιστοσύνη και υπομονή να αναμείνουμε να δούμε τι, τι θα γίνει. Και σε σχέση με μια χώρα που ενδιαφέρεται για τους Τσιγκάνους, τότε η Ουγγαρία ήταν μια τέτοια χώρα, άσχετα ποιο ήταν στην κυβέρνηση. Ας μην παίρνουμε μεμονωμένες περιπτώσεις τώρα. Σε όλες μας τις χώρες έχουμε έχουμε ριζοσπαστικές ακραίες τάσεις. Σε κάποιες χώρες περισσότερο, σε κάποιες άλλες λιγότερο. Σε κάποιες χώρες είναι η Ρωμά, η Τσιγκάνη στόχος, σε άλλες η Μωαμεθανή, η, ε, το Ισλάμ, ε, η Αλόδοξη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν, να μην καταδικάζουμε συλλήβδιν. Και τώρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που άκουσα από εσά και από άλλους προηγούμενα, αν η κυβέρνηση θέλει να μεριμνήσει στην Ουγγαρία τα προβλήματα των Τσιγκάνων να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει με θετικό τρόπο, με καλή παιδεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, τότε καλό είναι αυτό. Ο αντισημιτισμός δεν είναι θέμα εξειδικευμένα ουγγρικό, είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα, αφορά όλες μας τις χώρες ο αντισημιτισμός. Α το δούμε αυτό και να το συνειδητοποιήσουμε και α μην δακτυλοδεικτούμε και καταγγέλουμε τους άλλους. Ε, υπάρχουν τάσεις εδώ που λόγω της Γερμανίας και του φρικαλαίου παρελθόντο τη ε, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Αλλά και σε άλλε χώρε υπάρχουν ε, συναφείς τάσει. Α μην απλοποιούμε τα πράγματα λέγοντας ότι τώρα επειδή έχει την Προεδρία η Ουγγαρία υφίσταται αυτές τις επικρίσεις και επιθέσεις. Αυτά ήθελα να πω για να τα εκφράσω με ειλικρίνεια και ελεύθερα. Πρέπει πιο σφαιρικά και πιο συνολικά να τα δούμε τα πράγματα. Πρέπει να δίνουμε συνέχεια όμως σε αυτά τα θέματα. Τα ανέφερε αυτά ο κύριος Καβαντά, έδωσε συνέχεια η κυρία Τρούπερ. Εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δούμε τι κάνει η κυβέρνηση πραγματικά και ποιες είναι οι προθέσεις της. Και είμαστε βέβαιοι ότι οι μορφωμένοι πολιτισμένοι άνθρωποι σε αυτή την κυβέρνηση θα βρουν τη σωστή οδό. Για την πολιτισμική πορεία μιας κυβέρνησης σε μια χώρα, όταν κλείνει ένα θέατρο, αν ενδιαφερόμαστε και όταν ενδιαφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, τότε νομίζω ότι πάμε ένα βήμα πέρα από τα εσκαμμένα. Θέλουμε να λειτουργούν τα θέατρα και κινηματογράφοι. Αν κάπου όμω για κάποιου λόγου, ίσω και για του εσφαλμένου λόγου, λανθασμένου λόγου, υπάρχει εξοικονόμηση όσον αφορά τα κονδύλια για τον πολιτισμό. Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Παντού συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό όταν δακτυλοδεικτούμε κάποιον και καταγγέλνουμε, καταγγέλουμε να ξέρουμε ότι αυτό θα επιστρέψει σε εμά ω κατηγορία και καταγγελία. Λοιπόν, σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ Πολιτισμού. Μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο συνάδελφο που θα παρέμβει τώρα. Ευχαριστώ. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν ήρεμα παρακαλώ και όσοι θέλουν να συζητήσουν επίσης. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε για την νεολαία, για την νεότητα ορισμένα πράγματα, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε Φάκολα, θέλουμε να συζητήσουμε για τα θέματα της νεολαίας, της νεότητας. Χαιρόμαστε που μπορούμε να έχουμε μια τοποθέτηση που από εκείνον τον Υπουργό που είναι αρμόδιος στην Προεδρία την Ουγγρική θα μας μιλήσει για το πολιετές πρόγραμμα για τη νεότητα και την νεολαία. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να μας ε, δώσετε ελπίδες ότι υπάρχουν νέες ιδέες ε, και δυνατότητες που από κοινού μπορούν να προαχθούν. Κύριε Σόλτες, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε αυτό το μάθημα Ουγγρικής. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Θα πρέπει να σας κάνω μία σύντομη ανασκόπηση των προτεραιοτήτων και σχεδίων της Ουγγρικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμεινο. Το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας ε, συνδυάζεται με τις αποφάσεις και προγράμματα της ε, Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και επίσης με τις πολιτικές αποφάσεις που αποτελούν την βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την νεολαία. Ε, θα ήθελα κάποια λεπτά προσοχή, την προσοχή σας για να κάνω μια σύντομη ανασκόπηση λοιπόν των προτεραιοτήτων μας για τους έξι μήνες που ξεκινάνε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Νεολαίας ε, δράζεται σε τρεις κύριους πυλώνες. Πρώτον, το νέο πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία από το 2010 μέχρι το 2018. Αυτή είναι η περίοδος που καλύπτεται. Και εδώ έχουμε 8 στόχους κλειδιά που επικαλύπτονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σας. Εκπαίδευση και κατάρτιση είναι οι σημαντικότεροι στόχοι. Υπάρχουν άλλοι δύο στόχοι που σχετίζονται με την πολιτική σχετικά με την νεολαία, συμμετοχή και εθελοντικές δραστηριότητες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία του, προγράμμα, του προγράμματος της Ουγγρικής Προεδρίας. Οι άλλοι στόχοι του πρώτου πυλώνα, μάλλον τους άλλους στόχους δεν θα τους αναλύσω λόγω έλλειψης χρόνου, μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα αν έχουμε χρόνο. Ο δεύτερος τώρα πυλώνας είναι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Νεολαία. Αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο αποτελεί μέρος της διαδικασίας της Λισαβόνας και ένα από τα κυριότερα μηνύματα είναι η συμμετοχή και εμπλοκή, ενεργός εμπλοκή των νέων στην πολιτική, στις καθημερινές ε, δραστηριότητες. Βλέπω αρκετούς νέους εδώ στην αίθουσα. Υπάρχουν νέοι που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα γενικά των νέων και της νεολαίας. Εκτός από τους τρεις πυλώνες πρέπει να αναφερθούμε και στο πρόγραμμα Youth on the Move, νεολαία εν κινήσει, που αντικαθιστά το σύμφωνο για την νεολαία. Άκουσα το πρωί αρκετέ ερωτήσει για τη χρηματοδότηση και το, ε, η νέη κινήση μπορεί να είναι μια από τι εμβληματικέ πρωτοβουλίε στη στρατηγική τη Ευρώπη 2020. Υπάρχουν αρκετέ εμβληματικέ πρωτοβουλίε στο έτο εκπαίδευση και στην πολιτική για την νεολαία και η ε, νέη εν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μας βοηθήσει να ε, προωθήσουμε αυτό το Τώρα, στο θέμα της κατάρτισης θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό απασχόλησης κυριότερα ανάμεσα στους νέους. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένας στους πέντε νέους ε, είναι άνεργοι, δεν έχουν μια θέση απασχόλησης. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Ιδιαίτερα αν το ε, εξετάσουμε υπό αυτό το πρίσμα. Είναι οι σημερινοί νέοι που θα πρέπει να υποστηρίξουν την ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα συστήματα, τα κοινωνικά, τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης στις επερχόμενες δεκαετίες. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε, έναν, σε ένα άλλο ρηξικέλευτο πρόγραμμα. Δηλαδή, έχει σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που ξεκινάει η Ουγγρική Προεδρία, διότι έχουμε μόλις ξεκινήσει, λανσάρει το έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων με πολλές προσδοκίες για τους νέους. Έντιμα μέλη, η τριανδία της Προεδρίας έχει ένα κοινό πρόγραμμα και σε αυτό το πρόγραμμα η Ουγγρική Προεδρία θέλει να κτίσει στα επιτεύγματα της Βελικής και Ισπανικής Προεδρίας και ε, σε αυτή την τριαδρία θα θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως στην απασχόληση των νέων. Η Ισπανική Προεδρία εστίασε την προσοχή της στην κοινωνική συμπερίληψη. Ήταν η πρώτη παρελθόν ένα προτεραιότητα. Κατά το εξάμεινο της Βελικής Προεδρίας η πρώτη προτεραιότητα ήταν η απασχόληση των νέων και τώρα στην, το τρίτο εξάμεινο της Τριανδρίας είναι, το θέμα μας είναι η συμμετοχή των νέων. Συμμετοχή και ιδιαίτερα στο θέμα της απασχόλησης των νέων. Τι σημαίνει συμμετοχή. Σημαίνει, σημαίνει ενεργός πολιτότητα, συμμετοχή στα πολιτικά, ε, συμμετοχή στην δημόσια ζωή, συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι εξίσου σημαντικό, όπως το έχω ήδη αναφέρει, να δώσουμε την ε, ευκαιρία στους νέους να συμμετέχουν στα δημόσια, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί οι εντάσεις που έχουμε αισθανθεί και ακόμη και σήμερα ε, εξομαλύνονται πιο εύκολα αυτές οι εντάσεις όταν οι νέοι έχουν την ευκαιρία να τα συζητήσουν γιατί ε, πολλές φορές ε, υπάρχει καλύτερη αλληλοκατανόηση ανάμεσά τους. Είναι γι' αυτό που η συμμετοχή των νέων στα πολιτικά δρόμενα είναι πολύ σημαντική και μπορεί να έχει πολλά ωφέλη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις εθελοντικές δραστηριότητες. Οι εθελοντές συναντώνται πιο συχνά στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς δεν έχουμε τόσες εμπειρίες με τον εθελοντισμό στην Ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Αλλά αν θέλει κανείς να πετύχει, ε, θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα σε κάθε ξεχωριστό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει και όχι μόνο όταν μιλάμε για το ευρωπαϊκό έτος ε, του εθελοντισμού θέλουμε και τη συμμετοχή μη ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τρίτες χώρες διότι με τη μελλοντική διεύρυνση οι νέοι, οι σημερινοί νέοι σε αυτές τις χώρες θα είναι οι αυριανοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Προεδρία κατά την συνεδρίαση ε, που έγινε τον Μάιο ε, θα ήθελε να εγκρίνει ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου στο θέμα των νέων. Θα ήθελα ε, να πω κάτι για τον δομημένο διάλογο. Είναι ένας άλλος ε, τομέας προτεραιότητας για μας και στενά συνδεδεμένος με την απασχόληση των νέων. Όταν συμφωνήσαμε με τους Ισπανούς και Βέλγους συναδέλφους να το θέσουμε ως προτεραιότητα, θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας από τη βάση στην κοροφή. Θέλαμε να ξεκινήσουμε από το επίπεδο το βασικό, από τη βάση και να εμπλέξουμε τους νέους. Οι νέοι να προτείνουν τις ιδέες τους, τις επιθυμίες τους, τις προτάσεις τους και ε, θέλουμε να διοχετεύσουμε αυτές τις προτάσεις και ιδέες ε, στους ηθήνοντες ε, πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η χάραξη πολιτικής που έχουμε εμείς κατά νου. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας καλέσω στο συνέδριο Ευρωπαϊκής Νεολαίας ε, από τις 2 στις 4 Μαρτίου στη Βουδαπέστη, λίγο έξω από τη Βουδαπέστη, στο Γκέντελε, στην πόλη του Γκέντελε. Σε αυτό το συνέδριο θα συμμετέχουν όλοι οι σημαντική συμμετοχή στον τομέα της πολιτικής για τους νέους και επίσης ελπίζουμε να εγκριθούν συμπεράσματα Συμβουλίου τον Μάιο. Αυτά τα συμπεράσματα θα είναι πολιτικής φύσεως και θα καθορίζουν τις προτεραιότητες για τις επόμενες ε, προεδρίες στην Πολωνική και την ε, Δανέζικη. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κλείσω την παρουσίασή μου. Ε, μου έχει υποδείξει η Πρόεδρος ότι θα πρέπει να συντομεύω. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν όχι μόνο στην Ουγγαρία. Θα υπάρχουν και παρόμοια γεγονότα και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, στις Βρυξέλλες για παράδειγμα ή επίσης ε, το έτος ε, νεολαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Είναι όλα αυτά τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα που εξυπηρετούν στο να αυξάνουν τη συμμετοχή και εμπλοκή των νέων στα δημόσια, στην ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία, στα πολιτικά δρόμενα και είναι ιδιαίτερα σε αυτό που θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην Ουγγρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς τώρα πιέζει πολύ ο χρόνος και αυτό οφείλεται στον πολύ χρόνο με τον οποίο συζητούσαμε με τον Υπουργό Πολιτισμού. Όχι ότι έχουμε λιγότερο ενδιαφέρον για το δικό σας πεδίο, αλλά πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι. Ο συνάδελφος Φίσας και μετά ο συνάδελφος Τάκουλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την τοποθέτησή σας. Αυτή τη στιγμή, κυρία Βασιλείου, υποδέχεται την διακομματική ομάδα για την νεολαία αυτής της Ευρωβουλής είχε υπάρξει πρόσκληση να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Είμαστε εδώ στην Ευρωβουλή για να ακούσουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Έχουμε πολλά θέματα που συνδέονται με την νεότητα, με την νεολαία. Για τα όσα αναφέρθηκε για την πολιτική συμμετοχή των νέων είναι πολύ σημαντικά και εδώ και πολλά χρόνια και με το θάνατο του Φράγκο στην Ισπανία, εκείνη τη χρονική συγκυρία υπήρχε ενθουσιασμός όσον αφορά τη νεολαία, τους νέους, γενικά και στην Ευρώπη για τα πολιτικά θέματα. Πιστεύω ότι είναι και είναι μια προσωπική άποψη ότι επίσης πρέπει να αποφύγουμε την επαγγελματοποίηση, επαγγελματική εμπλοκή των νέων χωρίς να υπάρχει μια επαρκής ε, ε ακαδημαϊκή ε, θα έλεγα από πλευράς ε, παιδείας και εκπαίδευσης ε, δυνατότητα τα μάθησης. Και εδώ θα ήθελα να σχολιάσω δύο θέματα. Κάνατε λόγο για την εθελοντική εργασία και συμμετοχή. Τι αναμένετε για το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντών. Ποιες προσδοκίες έχετε. Και Κάπως αν μπορείτε να αναπτύξετε το θέμα για τις, ε, τη νεότητα. Το πρόγραμμα Έρασμος, ε, αν μπορείτε να το ε, αναφέρετε, έχει κάνει πολλά πράγματα για τους νέους, πολλά περισσότερα από πολλές συνθήκες και άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε Τάκουλα, τώρα πολύ σύντομα, παρακαλώ εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για μια πολύ καλή έκθεση, εισήγηση από πλευρά του. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας έχουμε μια πολύ καλή στάση, προσέγγιση, τοποθέτηση. Θέλετε πολλά να ε, πετύχετε. Αν θέλετε όλα αυτά να περάσουν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και το καταφέρετε, αυτή η Ουγγρική Προεδρία θα στεφθεί με επιτυχία. Και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρίας να γίνει αυτό, αλλά να τύχει και συνέχεια. Μία ερώτηση έχω. Κάνετε λόγο για την κοινωνική συνοχή και εκφράζετε και την ανησυχία σας για την ε, ανεργία των νέων που είναι πολύ υψηλή. Αληθεύει είναι γεγονός ότι 20% είναι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστιας εμβέλειας θέμα αυτό. Τώρα που έχουμε και την ελευθερία κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη, κατά κάποιο τρόπο αυτό θα πρέπει να θίγεται όπως ε, του αρμόζει κάνοντας λόγο για αυτή την πτυχή. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλά κράτη-μέλη το όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται, η επαγγελματική σταδιοδρομία των πολιτών επιμηκύνεται, υπάρχει ενθάρρυνση, προτρέπονται οι πολίτες να συνεχίσουν να εργάζονται στις, ε, ε, στους χώρους απασχόλησής τους. Και έχουμε και το φαινόμενο της μετανάστευσης από τρίτες χώρες προς την Ευρώπη. Είναι αξιοπερίεργη αυτή η εξίσωση. Ε, είναι υψηλό το ποσοστό ανεργία των νέων. Πολλοί θέλουν να συνταξιοδοτηθούν όταν φτάνουν το όριο συνταξιοδότηση. Του λένε όχι, να μείνετε στην απασχόλησή σα και πολλοί έρχονται ω μετανάστε να εργαστούν στην Ευρώπη επειδή υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό λοιπόν οπωσδήποτε των πολιτικών μα και των μέτρων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν αυτό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το καλύψουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Διότι εξαρτόμαστε από τους νέους για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να βρουν απασχόληση λοιπόν οι νέοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόρις παρακαλώ. Ε, chciałem też podziękować za to kompleksowe podejście i, i kontynuację działań prezydenta. Πολύ για αυτή την παρέμβαση που είσαι πλήρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ότι συνεχίζετε εσεί όλη την προσπάθεια που ξεκίνησαν οι προηγούμενε προεδρίε. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται για τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κίνα για την χρονιά που μα πέρασε, θα συνεχιστεί και δεύτερο ερώτημα όταν αφορά τους νέους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα υπάρχουν οικονομίες οι οποίες βασίζονται στο έρασμος. Υπάρχουν πολλοί φίλοι στην, στην οι οποίοι πρέπει να φύγουν από εκεί και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα πρόγραμμα για τους φοιτές της Βιελορουσίας και μπορούμε να τους βοηθήσουμε λόγω της πολιτικής καταστάσεως που υπάρχει σε αυτή τη χώρα και να θέλουν να σπουδάσουν δεν μπορούν να το επιτύχουν αυτό το πράγμα. Τι σκέφτεται γι' αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο ε, πολιτή. Ο κύριο Τέκιο, μία ερώτηση. Μόνο έχουμε μόνο πέντε λεπτά και ο Υπουργό πρέπει να απαντήσει. Παρακαλώ, κύριε Τέκιο. Μια μόνο ερώτηση, βέβαια. Είναι γνωστό ότι η Ουγγαρία αλλά και στην Ευρώπη, διότι έχουμε μια δημογραφική κρίση. Μπορεί να μην έχω λάθος όταν υποδεικνύω ότι η λύση μπορεί να έγκυται στο επίπεδο των νέων. Γνωρίζω, ε, Υπουργέ Σόλτες, ότι η Ουγγρική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία της οικογένειας και θα θέλει να αντιμετωπίσει αυτό την πρόκληση της δημογραφίας, των δημογραφικών δεδομένων. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι προθέσεις σας στην πολιτική για τους νέους, για την προστασία της οικογένειας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, των δημογραφικών προβλημάτων. Πρόεδρε, θα επιχειρήσω να παραμείνω στο χρόνο μου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι φυσικά η Επίτροπος Βασιλείου είχε ανταλλαγή απόψεων για τις εθελοντικές δραστηριότητες και αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Και είναι γι' αυτό που είχαμε πει ότι ο εθελοντισμός θα πρέπει να αποτελεί το θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο του Μαΐου. Θα πρέπει να αποτελεί θέμα στην ημερήσια. Όχι μόνο στην Ουγγαρία, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε σχόλια από κοινωνιολόγους και από μελέτες που, υποδεικνύουν ότι αν εμπλακούν οι νέοι σε θελοντικές δραστηριότητες, αν συμμετέχουν σε κοινωνικά ιδρύματα, ιδρύματα περίθαλψης, θεραπείας, φροντίδας αναπήρων, αν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εργασίες, τότε σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους ε, θα έχουν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία και στάση, θα είναι πιο ανοιχτή, θα είναι πιο ανεκτική απέναντι σε αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Αυτό το έτος του εθελοντισμού, σε αυτό το έτος του εθελοντισμού αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Γιατί υπάρχουν πολλά άτομα με στην Ευρώπη. Ε, μιλάμε για τεράστιους αριθμούς ανθρώπων και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ενισχύοντας την αλληλεγγύη στην κοινωνία και ε, μπορεί αυτό να ξεκινήσει από τους νέους. Για να απαντήσω στον κύριο Τάκλα για τη ε, σχετικά με την κοινωνική συνοχή και τους νέους και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Το πρόγραμμα που παρουσίασα και που ε, ενσωματώνεται σε μια σειρά προγραμμάτων ε, διάρκειας 6-7 ετών ελπίζουμε να μπορεί να αποδώσει κάποια καθήκοντα που θα ε, υποβληθούν ε, στην Επιτροπή την Άνοιξη για να εντοπίσουμε τα πιο φλέγοντα ε, θέματα στη ζωή των νέων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων απασχόλησης. Έχετε απόλυτο δίκαιο όπου λέτε ότι εκτός από την απασχόληση πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την έλλειψη εργασίας. Είναι θέμα επαγγελματική κατάρτισης και εκπαίδευσης για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά σχετίζεται και με τις πολιτικές, πολιτικές ε, νεολαίας και είναι συναφές όχι μόνο με τα ε, δικές σας αρμοδιότητες αλλά και τις αρμοδιότητες άλλων ε, επιτροπών στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή προσέγγιση αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Τώρα, απάντηση στον κύριο Μπόρις. Ε, το έτος νεολαίας Ευρώπης Κίνας. Μπορεί να γνωρίζετε πόσο μεγάλη οικονομική ε, επιτυχία και μεγάλη εξέλιξη έχει θεωρηθεί αυτό στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Πριν από δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τελετή εδώ στις Βρυξέλλες και τονίστηκαν τρεις πτυχέ από τους κύριους ομιλητές. Πρώτον, η πολιτιστική συνεργασία που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις αξίες μας και να τις αποδεχθούμε. Ο άλλος τομέας είναι η συνεργασία στην εκπαίδευση και ο τρίτος είναι η οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Οι πρώτοι δύο είναι εξίσου σημαντικοί με την οικονομική συνεργασία, διότι ο πολιτισμός είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα και που μας ενώνει. Η οικονομική συνεργασία μπορεί να μας βοηθήσει εμάς ε, και μας τους Ευρωπαίους και τους νέους στην Ευρώπη και μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενισχύσει την αγορά εργασίας. Χωρίς αγορά εργασίας δεν μπορεί κανείς να λύσει τα προβλήματα των νέων γενικώς θα πρέπει να βελτιωθούν η θέση στην αγορά εργασία και να βοηθήσουμε τους νέους να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία. σχετικά με τους Ρώσους και την κινητικό, η κινητικότητα των νέων είναι ένα μείζον θέμα. Ε, λυπάμαι πραγματικά που ε, υπάρχουν χώρες γείτονες Ευρωπαϊκής, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τόσα προβλήματα ε, και ε, ανάμεσα στους νέους και είναι κρίμα που η Λευκορωσία έχει τέτοια προβλήματα. Θα πρέπει να ανορχιστρώσουμε τη θέση μας με την ρωσική ηγεσία επίσης. Κινητικότητα των φοιτητών και προγράμματα τέτοια κινητικότητα μπορούν να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε τις ε, προοπτικές ε, των λευκορώσων φοιτητών και των νέων γενικώ. Είναι δύσκολο να δώσω μια σύντομη απάντηση στην ερώτηση του κ. Τόκερς, διότι οι πολιτικές για την οικογένεια και για τους νέους ε, είναι αλληλένδετες και καθορίζουν το μέλλον της Ευρώπης η Ευρώπη θέλει να παραμείνει ισχυρή και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας, τόσο το πολιτιστικό, το οικονομικό και το κοινωνικό πλαίσιο και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε πολιτικές για τους νέους και την οικογένεια και το τελευταίο εξάμεινο η γουρική κυβέρνηση προσπάθησε να αναπτύξει πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εκβάσεις. Ε, Μαθαίνουμε από άλλες χώρες φυσικά, από χώρες της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, από τη Γερμανία, την Γαλλία, αλλά μπορούμε πάντα να κάνουμε ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών ανάμεσά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Πάντα συμβαίνει στην αρχή, κατά τη διάρκεια μια προεδρία, να θεωρεί κανεί ότι του επόμενου έξι μήνε θα γίνουν πάρα πολλά και θα επιτευχθούν πάρα πολλά. Ξέρουμε όμω όλοι ότι πάντα μικρά βήματα μπορεί να είναι αυτή η πορεία. Αυτά όμω προστίθενται και στα επόμενα τη Πολωνική Προεδρία και ακολουθούν τα βήματα τη Βέλγικη Προεδρία. Είναι κοινοτικό το εγχείρημα. Εκεί όπου μα χρειάζεστε θα σα υποστηρίξουμε με προθυμία ιδιαίτερα ευχάριστα. Και ελπίζουμε φυσικά ότι κατά διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας θα τεθεί η τροχιά, θα χαραχθεί πορεία για προγράμματα και για την πρικοδότησή τους και έτσι για τον πολιτισμό, για τους νέους θα χρειάζονται κονδύλια. Όλοι μας πήραμε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε και πάλι εσά. ευχαριστούμε τους συναδέλφους που άντεξαν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και συνόδευσαν τη δουλειά μα με ερωτήσει. Κερδίσαμε μια επισκόπηση του έργου της Ουγγρικής Προεδρίας και ευχόμαστε για άλλη μια φορά αυτό το νομοθέτημα για τα μέσα ενημέρωσης να μην επισκιάζει τα πάντα στο μέλλον και επιτέλους οι αναγκαίες προσαρμογές να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και έτσι θα μπορούμε να ε, στρεφόμαστε με εμπιστοσύνη σε αυτή την Ουγγρική κυβέρνηση που θέλει να είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα και ελπίζουμε δεν θα μας απογοητεύσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απολύεστε τώρα κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Ο κύριος Ιβαν δεν θα μπορέσει τώρα να κάνει την παρουσίασή του. Δεν θα τα καταφέρουμε. Παρακαλώ αν γίνεται στις 5 η ώρα να είναι παρόν. Στις 5 η ώρα μετά από τη συζήτηση με την κυρία Ρέντινγκ θα έρθει το θέμα, η σειρά του θέματος του δικού σας. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και λίγη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ. Γεια σας.